Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Καλησπέρα κύριε και συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ήτρα. Καταρχήν, έγκριση της ημερήσιας διάταξης, δεν υπάρχουν σχόλια, οπότε θεωρούμε την ημερήσια διάταξη εγκεκριμένη χωρίς καμία μεταβολή. Και Πάμε και τα διάφορα ούτω ή άλλω στην ημερήσια διάταξη, οπότε είναι πολύ εύκολο να προσθέσετε κάτι. Δεν υπάρχουν σχόλια. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο, ανακοινώσει του Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση από την πλευρά μου και πιο σημαντική. Τα σημεία 5 και 6 τη ημερήσια διάταξη θα αλλάξουν σειρά μεταξύ του. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πάτρικ και Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας τη Αεροπορίας και μετά ο συνάδελφό μα ο κύριος Λάγκεν θα κάνει την ε, παρουσίαση σε ό,τι αφορά το σύστημα εμπορία εκπομπών, το ETS, ε, στον, ε, στην αεροπορία. Και αυτό λόγω της συζήτηση που θα γίνει στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και λόγω τη οποία ο συνάδελφο Λάγκεν δεν θα μπορεί να παρευρίσκεται στη συνεδρίασή μα την ε, προβλεπόμενη ώρα. Αυτό είναι ο λόγο δηλαδή που άλλαξε η σειρά αυτών των δύο σημείων 5 και 6 τη ημερησία διάταξη. Τώρα, μετά, ε, ακρόαση επιτρόπου. 15 λοιπόν Μαΐου του 2017 ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια επιστολή με την οποία ενημέρωνε το Κοινοβούλιο ως προς τον ορισμό της κυρίας Μαρία Γκάμπριελ ως οριστή σας επιτρόπου. Σύμφωνα λοιπόν με τους στον κανονισμό μας ε, οι ακροάσεις ε, των ε, επιτρόπων που έχουν ήδη οριστεί διοργανώνονται από τη διάσκεψη των Προέδρων. Ωστόσο, εμείς ως Επιτροπή Ήτρε θα μπορούσαμε να οριστούμε η αρμόδια επιτροπή για αυτή τη διοργάνωση. Οπότε, ο Πρόεδρος και οι συντονιστές κάθε συναφούς επιτροπής, κοινοβουλευτικής επιτροπής, είναι αρμόδιοι για τις ε, επιμέρους λεπτομέρειες της διοργάνωσης δηλαδή της ακρόασης. Και αν ανατεθεί στην ε, Επιτροπή Ήτρε αυτή η ακρόαση και είναι σχεδόν σίγουρο ότι αυτό θα γίνει, δηλαδή ότι θα είναι δική μας ευθύνη, τότε θα μπορούσε να λάβει χώρα μια ακρόαση με την οστήσα επίτροπο πριν από ε, το θερινό διάλειμμα θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Όπως γνωρίζετε, με τον Επίτροπο Έτινιο έχουμε κοινή ευθύνη για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και από κοινού με τους ε, συναδέλφους από την Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Παιδείας. Οπότε, ουσιαστικά, η ίδια διαδικασία θα είναι όπως αυτή που είχε λάβει χώρα την τελευταία φορά. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τώρα τις ανακοινώσεις από την πλευρά μου. Οπότε περνάμε στο σημείο 3 τη σημερινή σα διάταξη, δηλαδή παρουσίαση τη ειδική έκθεση του Ελεγχτικού συνεδρίου σε σχέση με τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον παροπλισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων, ανταλλαγή εδώ απόψεων με τον Phil Βιν Owen, μέλος του Ελεγχτικού συνεδρίου. Σα καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Owen, και χαιρόμαστε πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ για να ακούσουμε την παρουσίαση αυτή. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα αυτό για μας, ο παροπλισμός των πυρηνικών εγκαταστάσεων και πριν από 10 χρόνια ήταν ε, ιδιαίτερος δημοφιλές ο ζήτημα. Τώρα λοιπόν ε, έχει βγει λίγο αν θέλετε από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τώρα θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο από εσά κύριε Ουόν που είστε επικεφαλής και του τμήματος 1 του Ελεκτικού συνεδρίου που είναι αρμόδιο για την βιώσιμη αξιοποίηση ε, και τις ε, βιώσιμες και τους βιώσιμους ε, πόρους να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Είστε απόφυτος του Πανεπιστημίου του Oxford αλλά και του London Business School και του Harvard, του Business School συγκεκριμένα, του Πανεπιστημίου του Harvard. Έχετε εργαστεί λοιπόν στο δημόσιο τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου, ειδικότερα ως Γενικός Διευθυντής του Ετμήματος Ενέργειας και Κλιματικής Μεταβολής. Πολύ ωραία τον Ιανουάριο λοιπόν του 2014 αναλάβατε καθήκοντα ως μέλος του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου. Ο λόγος λοιπόν είναι σε εσά κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την ευγενική παρουσίαση. Ε, καλησπέρα σε όλους. Ε, Σα ενημερώνω ότι η παρουσίαση μου συνοδεύεται από διαφάνειε εδώ στην οθόνη. Σα ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε να κάνουμε αυτή την ε, παρουσίαση. Έχω τον Πέκρο Ουλάντα, ο οποίο είναι και ελεγκτή και πρώην επιθεωρητής πυρηνικών εγκαταστάσεων, άρα εκεί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Η έκθεση αυτή δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2016 και την παρουσίασα στην Επιτροπή Ελέγχων των Προϋπολογισμών 19 Νοεμβρίου του 2016 και την παρουσίασα και στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου με τίτλο ε, «Παροπλισμός πυρηνικών εγκαταστάσεων. Μια νέα πρόκληση για την πυρηνική ασφάλεια». Ε, στις 6 Φεβρουαρίου έγινε αυτό το σεμινάριο και επίση ε, πιο πρόσφατα έκανα μια παρουσίαση στις 28 Απριλίου εδώ αυτή τη έκθεση στο Κοινοβούλιο της Λιθουανίας. Οπότε ζητώ συγγνώμη σε όσους ήδη έχουν παρακολουθήσει αυτή την έκθεση. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν το πώς έλαμε χώρα ο έλεγχος, τα πορίσματα και τις συστάσεις μας. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, αποτέλεσε συνέχεια μιας έκθεσης προηγούμενης που είχαμε συντάξει το 2011. Εκεί είχαμε εξετάσει ε, τις, ε, ή μάλλον εδώ εξετάσαμε τις εξελίξεις από εκείνη την έκθεση. Δηλαδή έχουμε καλύψει την περίοδο στον Απρίλιο του 2016. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν έχουν λάβει χώρα εδώ ε, κάποιες περαιτέρω εξελίξεις από τότε δηλαδή που ολοκληρώθηκε η σύνταξη αυτής της έκθεσης. Παρ' όλα αυτά όμως ε, θεωρούμε πως ε, ε, επί, λόγω του χαρακτήρα της διαδικασίας του παροπλισμού ε, πολλά από τα πορίσματά μας παραμένουν σε ισχύ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τους ε, πρώτης γενιάς ε, ε σοβιετικού τύπου πυρηνικούς ε, οι σχετικέ χώρε είχαν δεσμευτεί για την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση να του παροπλήσουν. Η Λιθουανία αντιμετώπισε ιδιαίτερη πρόκληση με αυτό, γιατί είναι σχετικά ε, μικρό κράτο μέλο, χωρί να έχει ιδιαίτερα ε, ανεπτυγμένο ενεργειακό τομέα και δύο ε, πυρηνικού αντιδραστήρε τύπου Τσενόμπιλ, του οποίου κλήθηκε να παροπλήσει, κάτι το οποίο δεν έχει λάβει χώρα στο παρελθόν. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε από το 1999 να παράσχει οικονομική υποστήριξη. Έως το 2020 η σχετική υποστήριξη προς αυτά τα τρία κράτη-μέλη για τον παροπλισμό θα έχει ανέλθει σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ με τη Λιθουανία να έχει λάβει περίπου το ίμιση αυτών των κοντιλίων. Εξετάσαμε λοιπόν την ε, πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την ε, τελευταία μας έκθεση και η διαφάνεια εδώ που βλέπετε ε, αναφέρει τη βασική ερώτηση ε, στην οποία βασίστηκε η έκθεση. Εμείς δεν καλύψαμε εδώ ζητήματα ε, συμμόρφωσης, ε, ζητήματα δημοσίων συμβάσεων ή ζητήματα ασφαλείας. Και σε καμία περίπτωση εδώ δεν θελήσαμε να ταχθούμε υπέρ ή κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας ή ως προς το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς έλαβε χώρα αυτός ο έλεγχος. Η δική μας ομάδα επισκέφθηκε αυτές τι τρεις εγκαταστάσεις. Εγώ προσωπικά επισκέφτηκα τις εγκαταστάσεις στη Λιθουανία και στη Βουλγαρία και συναντήθηκα και με εκπροσώπους της CBRD ε, και των σχετικών ε, εγκαταστάσεων όπως και με εκπροσώπους από το Γεωλογικό Αποθετήριο Πυρηνικών Αποβλήτων στην ε, Φιλανδία. Ποια είναι λοιπόν τα πορίσματα. Διαπιστώνουμε ότι έχει επιτευχθεί η πρόοδος από το 2011. Δηλαδή ο παροπλισμός ειδικότερα σε περιοχές ε, με χαμηλή ε, ε, ακτινοβολία έχει προχωρήσει αρκετά. Για παράδειγμα στους χώρους των τουρμπινών. Ωστόσο στους τομείς ή στους, στους χώρους εκείνους με υψηλή ραδιενέργεια δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά. Για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον παροπλισμό των ίδιων των αντιδραστήρων. Από εκεί και μετά τα χρηματοδοτικά προγράμματα για τον παροπλισμό δεν έχουν δημιουργήσει διαπιστώνουμε τα κατάλληλα κίνητρα για μια έγκαιρη και αποδοτική διαδικασία παροπλισμού. Έως τα τέλη του 2015 δεν είχαμε επιτύχει όλα τα ε, αναμενόμενα αποτελέσματα, όπως δηλαδή είχαν οριθεί από την Επιτροπή, ε, προκειμένου να θεωρηθεί πως η διαδικασία του παροπλισμού είναι μη αναστρέψιμη, irreversible η άδεια ε, για τις ε, μονάδες 3 και 4 ε, από τότε που συντάχθηκε η μελέτη μας έχει πλέον δοθεί στη Βουλγαρία οπότε εδώ θα έπρεπε να αλλάξει ένα από τα κουτιά που είδατε και να γίνει πράσινο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα απόλυτα να πούμε ότι ενώ υπάρχει πρόοδος κάποια από τα βασικά project, κάποια από τα βασικά έργα έχουν καθυστερήσει και εδώ αναφέρουμε κάποια στη Λιθουανία για παράδειγμα η ημερομηνία του παροπλισμού που ήταν, είχε προβληθεί ε, αρχικά ε, ε, για πολύ νωρίτερα, τελικά προβλέπεται πλέον το 2038. Επίσης, προκλήσεις παραμένουν και στα τρία κράτη-μέλη, ακριβώς λόγω των καθυστερήσεων σε ό,τι αφορά τα σχετικά έργα. Και ο διάλογος που έγινε σε ό,τι αφορά την οριστική απομάκρυνση από των πυρηνικών αποβλήτων βρίσκεται ακόμα στα πολύ αρχικά του στάδια. Οπότε, σε γενικές γραμμές, ε, Αντίσαμε το συμπέρασμα ότι το γενικό κόστος ε, για τον παροπλισμό αυτών των εγκαταστάσεων θα ανέλθει σε συνολικά 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και το χάσμα αν θέλετε ανάμεσα στις δαπάνε και το αναμενόμενο προϋπολογισμό ειδικότερα στη Λιθουανία, έχει ε, αυξηθεί κατά 1,5 ε, δισεκατομμύρια ευρώ στη Λιθουανία 25 ε, στην, ε, και 25 στη Βουλγαρία. Τώρα η συγχρηματοδότηση από την πλευρά των κρατών μελών παραμένει πολύ περιορισμένη ενώ το, ο αριθμός του προσωπικού είναι χαμηλός. Κάποια, κάποιο κόστος από αυτήν τις, τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αξιοποιηθεί για την καταβολή μισθών στο προσωπικό και όχι για τις δραστηριότητες του παροπλισμού. Από εκεί και μετά εδώ δεν έχουμε περιλάβει ε, το κόστος της οριστικής, τελικής δηλαδή απολύψης των αναλωμένων ε, καυσίμων και της απολύμανσης. Οπότε εδώ κάναμε και μια εκτίμηση του γενικού κόστους. Αν ε, δηλαδή εστιάσετε στην δεξιά στήλη, στην πρώτη γραμμή λοιπόν εκεί, πάνω δεξιά, βλέπουμε τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το συνολικό κόστος του παροπλισμού αυτών των εγκαταστάσεων. Όμως από εκεί και μετά προσθέτουμε την εκτίμηση σε ό,τι αφορά δηλαδή την απομάκρυνση ε, του, των αποβλήτων υψηλής ενέργειας. Και εδώ διπλασιάζεται δηλαδή με αυτό το κόστος. Ε, με, με την προσθήκη αυτή ακριβώς του κόστου τη απομάκρυνση σε συνολικά 11,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε πως η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά αυτές τις απορρίψει και η σχετική διαδικασία της εκ των προτέρων ερεσιμότητα ήταν ελλειπής. Δηλαδή το μελλοντικό κόστος για τον παροπλισμό και την οριστική απομάκρυνση των καυσίμων ε, δεν αναγνωρίζονται ως σχετικές διατάξεις, ούτε καταχωρίζονται με αυτόν τον τρόπο, ε, ε, με αποτέλεσμα βέβαια να μην υπάρχει κατάλληλη διαφάνεια και να μην αναλαμβάνουν τις ε, κατάλληλες ευθύνες οι αρμόδιες αρχές. Η Επιτροπή στην απάντηση που έδωσε στην έκθεσή μας μας ανέφερε ότι παραμένει δύο βασικά ορόσημα σε αυτές τις διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2016. Και πράγματι διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν Ειδικότερα πριν από δύο εβδομάδε ολοκληρώθηκε ένα σημαντικό ε, πρόγραμμα στι 15 Μαου συγκεκριμένα ε, στο πλαίσιο και τη εφαρμογή τη οδηγία για, ε, για τα πυρηνικά απόβλητα. Ποιε λοιπόν είναι οι συστάσει μα, θα τονίσω μόνο τέσσερι συστάσει σε ό,τι αφορά ειδικότερα την απόρριψη δηλαδή των πυρηνικών αποβλήτων υψηλή ραθιενέργεια και τη χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά τη σύσταση δύο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την οριστική απόρριψη. Λέμε λοιπόν εδώ ότι η Επιτροπή μαζί με όλα τα λεγόμενα κράτη-μέλη θα πρέπει να διερευνήσει τι αναλλακτικέ που έχει στη διάθεσή τη για την απόρριψη ε, των αναλωμένων καυσίμων και των αποβλήτων υψηλή ενέργεια, λαμβάνοντα υπόψη περιφερειακού και άλλε ευρωπαϊκού χαρακτήρα ε, λύσει, λαμβάνοντα βέβαια πάντα υπόψη την εσωτερική ασφάλεια, εξωτερική ασφάλεια και την, ε, μια σωστή σχέση κόστο αποτελέσματο. Ε, καλούμε από την Επιτροπή να επιληθεί αυτό το ζητήμα στο πλαίσιο τη πρώτη έκθεση που θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη οδηγία. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, κάναμε τρει συστάσει δηλαδή τη υπαριθμών 3, 4 και 5. Στη σύσταση 3 αναφέρουμε ότι τα τρία κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίσουν το ρόλο που τα ίδια θα πρέπει να παίξουν προκειμένου να διασφαλίσουν την ε, συμμόρφωση με την αρχή του ορυπαίνων πληρών και θα πρέπει κατά συνέπεια να αξιοποιήσουν εθνικά κονδύλια για να καλύψουν το κόστο του παροπλισμού αλλά και οριστική απόρριψη τόσο στο πλαίσιο τη ε, τρέχουσα χρηματοδοτικής περίοδου όσο και στο πλαίσιο τη μελλοντική. Στη σύσταση 4 αναφέρουμε πως η Επιτροπή θα πρέπει να αξιώσει υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της ε, ε περίοδου 2014-2020. Και στο, στην σύσταση 5 αναφέρουμε ότι ειδικά προγράμματα, πολιτιστικά προγράμματα ε, χρηματοδότηση του παραπλησμού στις τρεις ε, χώρες θα πρέπει να ε, πάυσουν, να τερματιστούν ε, έως το 2020. Και γιατί ακριβώς εννοούμε εδώ, και νομίζω πως έχει νόημα να διαβάσετε το σύνολο της έκθεσης. Λέμε ότι εάν υπάρχει εδώ μια σαφής ανάγκη για την αξιοποίηση ενωσιακών κονδυλίων ε, από το 2020 και μετά, θα μπορούσε αυτό να γίνει σε ένα ή σε περισσότερα από αυτά τα κράτη-μέλη. Αλλά οποιαδήποτε μελλοντική χρηματοδότηση αποφασιστεί, προταθεί δηλαδή από την Επιτροπή και συμφωνηθεί από του ε, συνομοθέτες, θα πρέπει να περιλαμβάνει και το σχετικό, τα, ζητήματα κινήτων και τα ζητήματα απομάκρυνσης των αποβλήτων. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ε, στο πλαίσιο αυτών των νέων προγραμμάτων και κατάλληλο επίπεδο συγχρηματοδότηση από την πλευρά των Είπαμε ότι ο ένας τρόπος ε, θα μπορούσε να είναι να υπάρξει ευρύτερη πρόσβαση στα κονδύλια των ευρωπαϊκών ε, διαχρονικών και επενδυτικών ταμείων έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση με τις ε, προϋποθέσεις που μόλις τώρα ανέφερα στο πλαίσιο της διαδικασίας παροπλισμού. Αυτά από την πλευρά μου και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ σαφής. Και μεστή. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα. Από το ΕΣΥΑΡΟ κ. Φόξ πρώτα. Πρώτα ευχαριστώ. Ευχαριστήσω τον κύριο Γουινόεν για την ξεκαθαρή παρουσίασή του. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ποιες είναι οι κοινωνικές ευθύνες της Ένωσης σε σχέση με αυτούς τους τρεις αντιδραστήρες γιατί από ό,τι είχα καταλάβει ήταν τμήμα του πακέτου προσχώρησης αυτών των τριών χωρών. Έχουμε όμως νομική υποχρέωση να γράψουμε μια λευκό επιταγή ή υπάρχει χρονοδιάγραμμα και προθεσμία. Θα ήθελα να μάθω πώς εμπλέκεται εδώ ο Ευρωπαίος φορολογούμενος σε σχέση με αυτούς τους τρεις αντιδραστήριες, να μας πείτε. Επίσης, είπατε ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έδινε τα σωστά κίνητρα Εμένα μου φαίνεται αυτό σαν να λέμε ότι να πάρτε εδώ ένα κορβανά με ευρωπαϊκά χρήματα και άρχισαν ευχαρίστως να τα δαπανούν οι τρεις χώρες αυτά τα χρήματα χωρίς να έχουμε εμείς κανένα έλεγχο. Για τη σύσταση 4, για την εθνική συγχρηματοδότηση, θα πρέπει να καθορίσουμε ξεκάθαρα στην απόφαση της Κομισιόν τις συνθήκες προς οποίες μπορεί να υπάρξει πλήρη χρηματοδότηση. Γιατί νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα είναι μάλλον εξαίρεση και όχι τόσο καλή εξαίρεση όσον αφορά τους φορολογούμενους. Μπορείτε λοιπόν να σχολιάσετε αυτά τα σημεία και ως ένα από τους ελεκτές και πρασπιστές του δημοσίου χρήματος να μας πείτε πώς έχουν δαπανηθεί τα χρήματα των φορολογουμένων μέχρι τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Από την ΚΟΕ, κύριος Κοκλίτσε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε την δαπάνη του δημοσίου χρήματος. Αλλά ίσως περισσότερο αυτό να αφορά αυτούς που διαπραγματεύτηκαν με αυτές τις χώρες μέλη, δηλαδή αυτούς που του, τις υποχρέωσαν να παροπλήσουν και να κλείσουν αυτούς τους τρεις αντιδραστήρες. Πρέπει λοιπόν αυτοί να βγουν μπροστά και να μας πούν ακριβώς τι πρόοδος έχει μεθεί σε αυτές τις χώρες, Βουλγαρία, Λιθουανία κτλ και να κάνουν και μια σύγκριση και να συγκρίνουν επίσης παρόμοιες διαδικασίες στη Γερμανία ας πούμε. Ναι, ίσως να μην ε, ε, είμαι σαφής. Συνεχίζω μιλητής. Θα πρέπει να συγκρίνουμε διαδικασίες παροπλισμού μεταξύ Γερμανίας οι οποίες εξελίσσονται βαθμια και γρήγορα παρά το γεγονό ότι η Γερμανία έχει κάποια προβλήματα με την προμήθεια ενέργεια και θα πρέπει να συγκρίνουμε λοιπόν αυτό με αυτά που συστήθηκαν από τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και την τρίτη χώρα. Και τι υποσχέσει δόθηκαν, α πούμε, στη Βουλγαρία. Γιατί υπήρχε στη Βουλγαρία ένα σχέδιο για νέες εγκαταστάσεις πυρηνικές αλλά μέχρι τώρα δεν έγινε ούτε μία αναφορά για το πώ η Βουλγαρία θα μπορούσε το Βιλ Μπέλενε και το Λέσκοφ. Τι γίνεται με τι επιπτώσει αυτών των δύο πυρηνικών, πυρηνικών εγκαταστάσεων στο κόστο του ηλεκτρικού ρεύματο. Και νομίζω το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για τι χώρε τη Βαλτική γιατί αποτελούν την κύρια πηγή τα πυρηνικά για την ενέργεια για την τροφοδότηση ενέργεια της χώρας. Οπότε θα ήθελα να μάθω ποιος είναι υπεύθυνο για αυτή την αποτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και ποια είναι η, η σύστασή σας, τι προτείνετε ακριβώ για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Thank you very much. Um, if may να αναφερθούμε και δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα. Υπάρχουν και άλλα πυρηνικά εργοστάσια τα οποία θα πρέπει να παραπληστούν στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επιχειρηματική ευκαιρία για κάποιους από εσά. Και υπάρχει άλλη μια ερώτηση. Είπατε ότι τα προγράμματα χρηματοδότησης της Ένωσης δεν δημιουργήσαν τα σωστά κίνητρα. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε την κατάσταση όταν δίδονται επαρκή κονδύλια ή τα σωστά κίνητρα για τον παραπλησμό. Και μετά, μια άλλη ερώτηση. Μετά από την τραγωδία της Φουκουσίμα, έχουμε εκπονήσει νέες κατευθυντές γραμμές στην Ευρώπη για την ασφάλεια στα πυρηνικά εργοστάσια. Όλα αυτά που έχουν γίνει λοιπόν μέχρι τώρα ήταν σύμφωνα με αυτούς τους νέους κανονισμούς ή όχι. Γιατί η διαδικασία του προπλισμού από ό,τι θυμάμαι ξεκίνησε πριν από το ατύχημα την τραγωδία στη Φουκουσίμα. Οπότε τίθεται το ερώτημα πώς εφαρμόστηκαν σε αυτή την περίπτωση οι νέοι κανονισμοί ασφαλείας. Να ρωτήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν έχουν κάποια σχόλια. Ο κύριος Γεράσιμος Τομάς, υποδιευθυντής από την Κοινή ενέργεια. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου για την έκθεση και την καλή δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου. Είχαμε θαυμάσια συνεργασία και υποδεχτήκαμε σχεδόν όλες τις συστάσεις. Να πω δύο πράγματα σε σχέση με αυτά που συνέβησαν από τότε που άρχισε ο έλεγχος. Καταρχάς, για τις συστάσεις. Εδώ έχουμε τα προγράμματα παροπλισμού για αυτές τις τρεις ε, χώρες συγκεκριμένα και κάποιες άλλες συστάσεις είναι γενικότερες. Κάποιες αφορούν αυτές τις τρεις, άλλες γενικότερες. Για αυτά τα προγράμματα η Κομισιόν έχει ολοκληρώσει και εσωτερικές και εξωτερικές μελέτες που επιβεβαιώνουν το ότι οι αξιολογήσεις εκ των προτέρων αλλά και εκ των υστέρων τηρούν τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις τους χρηματοοικονομικούς. Όταν έχει γίνει ο έλεγχος δεν είχαμε τεκμηριώσει όλα αυτά τα στοιχεία δεόντως, αλλά τώρα έχουν τεκμηριωθεί τα πάντα από πέρσι και το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει χρηματοοικονομικό κενό για το τωρινό πλαίσιο και τα κόστη, οι υπολογισμοί κόστους είναι σωστά μετά τον έλεγχο δηλαδή. Δεύτερον, η Κομισιόν ενίσχυσε την διαφάνεια αυτών των τριών προγραμμάτων και δημοσίευσε μια αιτήσια έκθεση που μεταβίβασε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και αυτή του 16 θα είναι έτοιμη πριν τις διακοπές της καλοκαιρινές και θα δώσει περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, η δουλειά μας και η στόχευσή μας ήταν να βελτιώσουμε την ασφάλεια και αυτό ως τμήμα των συστάσεων πέρα δηλαδή των κυρίων σημείων παρέμβασής μας και επικεντρωθήκαμε λοιπόν σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ασφαλίσουμε μέχρι το 2020 το αμετάκλητο της διαδικασίας αυτής παροπλισμού και για την περίπτωση της Λιθουανίας είχαμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα οι Λιθουανικές αρχές αντιμετώπισαν προσφυγές, είχαμε καθυστερήσεις. Τώρα βρισκόμαστε στην ε, τελική φάση της διαδικασίας απομάκρυνση από το πυρηνικό καύσιμο. Πάντως όλες οι χώρες έχουν μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τη νέα οδηγία για τα πυρηνικά απόβλητα και έχουν καταθέσει έγκαιρα εθνικά προγράμματα και εθνικές εκθέσεις έχουν ανταποκριθεί στα ερωτήματα και στα αιτήματα της Κομισιόν αυτό και για τις τρεις χώρες. Νομίζω ότι πραγματικά προχωράνε, έχουν προχωρήσει πολύ με το θέμα της διαφάνειας και, της, και του συμβασμού με τη δευτερεύουσα απορρέουσα νομοθεσία. Μετά, για τη χρηματοδότηση. Έχουμε εδώ μια αύξηση μετά από τις συστάσεις του Ελεκτρικού Συνεδρίου και με χαρά να σας πω ότι η Σλοβακία ας πούμε, η χρηματοδότηση έχει αυξηθεί κατά 4,5% από το 2015 στο 2016. Στη Λιθουανία είχαμε μια αύξηση από το 17,6% το 2015 στο 20% το 2016. Οπότε, όπως βλέπετε, έχουμε συνεχή σταθερή αύξηση εκεί όπου ήταν χαμηλότερη η χρηματοδότηση. Μετά το 2020 δεν έχουμε κάποια νομική υποχρέωση να συνεχίσουμε να παράσχουμε στήριξη σε αυτά τα τρία προγράμματα. Έχουμε κάνει μια διάμεση αξιολόγηση και μια αξιολόγηση αντικτύπου για να δούμε ακριβώς αν θα χρειαστεί περισσότερη αρρωγή αλλά προσπαθήσαμε να πετύχουμε ότι εν λόγω χώρες θα έχουν επαρκή πόρους και χρηματοδότηση μετά τη συνέχιση του προγράμματος, δηλαδή το 2020, αν χρειαστούν. Και τέλος, όπως ανέφερε και το μέλος του συνεδρίου, πριν δύο εβδομάδες δημοσιεύσαμε την έκθεσή μας προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση των αποβλήτων όσον αφορά όλη την Ένωση και μιλήσαμε συγκεκριμένα για τα πυρηνικά καύσιμα. Τονίσαμε τις αλλαγές, Υπογραμμίσαμε το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση και διαφάνεια στη χρηματοδότηση και η κατάλληλη δικασία διάθεση των αποβλήτων. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση. Την δημοσιεύουμε κάθε τρία χρόνια και μα επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο να ασκήσουμε πίεση και να στοχεύσουμε στα προβλήματα σε κάθε χώρα μέλος και προσβλέπω βεβαίω την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτή την έκθεση, η οποία θα αφορά όλε τι χώρε μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Κύριε Φέγκρα, παρακαλώ, αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ναι, μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Δεν κατάλαβα τη σύσταση 2α. Βλέπω εδώ διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Η κάθε χώρα να αναλάβει τις ευθύνες της για την διάθεση των πυρηνικών αποβλήτων. Αυτό έχει το πλεονέκτημα της αφούς απόδοσης ευθύνης. Ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι η χώρα μπορεί να μην βρίσκεται στην ιδανική τοποθεσία. Το δεύτερο είναι να βρούμε έναν άλλο τόπο κάπου αλλού στην Ευρώπη. Αυτό έχει το μειονέκτημα ότι ξαφνικά η Κομισιόν είναι αρμόδια, το οποίο μπορεί και να σημαίνει ότι κανείς δεν είναι αρμόδιος, αλλά μπορεί όντως εν τέλει να βρούμε μια καλή τοποθεσία. Και η τρίτη εναλλακτική λύση είναι να εξεύρουμε μια ακόμα πιο κατάλληλη τοποθεσία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω, για παράδειγμα, ότι η Αυστραλία ενδέχεται να ενδιαφέρεται. Συνεπώς, το ερώτημα μου είναι το εξής. Ωραία, υποβάλλετε κάποιε συστάσει, αλλά μεταξύ των τριών διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων, εσεί τι προτείνετε τελικώ. Να σας πω, στην σύσταση του ελεγκτικού συνεδρίου, και ας το εξηγήσει το ελεγκτικό συνεδρίο, να μας πούν τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Εμείς πάντως δεχθήκαμε να ξεκινήσει μια συζήτηση. είναι ότι η σχετική οδηγία για τα αρτηνικά απόλυτα είναι σαφέστατη. Η χώρα μέλος και η επιχείρηση η οποία χειρίζεται τα ρεδινεργά απόλυτα έχουν την ευθύνη. Η οδηγία επίσης υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την τελική διάθεση. Δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν τη σχετική απόφαση. Εν τούτης, δεν αποκλείεται να εξευρεθούν σε εργατικές λύσεις ανά την Ευρώπη. Μάλιστα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη, παρατρύνουμε τα κράτη-μέλη να συζητήσουν ε, ενδεχομένες περιφερειακού χαρακτήρα λύσεις. Την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πυρηνικής Ενέργειας στην Πράγα φιλοξένησε ένα πάνελ με ομιλητέ από κράτη-μέλη, εμπειρογνώμονε και συζήτησαμε τα υπέρ και τα κατά τη κάθε Επίση, εξετάσαμε και το άλλο ενδεχόμενο. Με βάση το δεδομένο ότι τα ενεργά απόβλητα δεν είναι προνόμιο ούτως υπήν των χωρών που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από σχάσιμο υλικό. Όχι. Έχουμε ραδιοσότοπα για ιατρικέ χρήσει. Ε, θέλω να πω, ραδιενεργά απόβλητα παράγουν όλες λίγο πολύ οι χώρες. Συνεπώς, η εξέβρεση του κατάλληλου χώρου τελικής αναπόθεση είναι μια σημαντική υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο χειριστής ή η εταιρεία η οποία χειρίζεται τα υλικά έχει την τελική ευθύνη. Ακόμα και αν ε, υπάρχουν και μεσολογούν δεν αποκλείεται από την νομοθεσία μας δύο κρατημέλη να δεθούν να επιμεριστεί η παραγωγοί. επισης δεν αποκλειεται απο την νομοθεσια μας δυο κρατημελη να δεθουν να επιμεριστει η ευθυνη της τελικής διάθεσης των ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ των δύο χωρών. Έχει ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ εμπειρογνωμών στα κρατημέλη και μάλιστα κάποιοι εμπειρογνώμων στην συνεδρίαση της περισσότερης εβδομάδας εξέφρασαν σχετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, είναι ανοιχτή ως προς την εξέβρεση κοινών, επαναλαμβάνω, λύσεων μεταξύ χωρών μιλών. Ε, δεν συζητήσαμε πάντως καθόλου την πιθανότητα να αποσταλούν τα απόβλητα εκτός Ευρώπης. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριος Owen ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου τώρα θα σχολιάσει και θα απαντήσει τα, τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Πρόεδρε, πολλές ερωτήσεις θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά και ίσως να συμπληρώσω με κάποιες παρατηρήσεις αν και η Κομισιόν διαπίνησε κάποια από τα ερωτήματα. Κύριε Φόξ, ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας ως προς το κατά πόσον έχει νομική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους τρεις δηλαδή αντιδραστήρες, ο Γεράσιμος σας έδωσε πολύ σαφή απάντηση. Η Κομισιόν δεν θεωρεί ότι έχει κάποια ε, ευθύνη πέραν του 2020 και να συμπληρώσω ότι η μελέτη αξιολόγηση επιπτώσεων του 2011 λέει ότι δεν σκοπεύει η Κομισιόν να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το πράγμα μετά από το 2020. Και αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Θα έλεγα επίσης εκ μέρους των συναδέλφων από την Λιθουανία και το είπα αυτό στην ομιλία μου πρόκειται για ένα μικρό, πολύ μικρό κράτος μέλος με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να αποσυναμολογήσει να παροπλήσει έναν ε, αντιδραστήριο τύπου Τσενομπίλ. Στο άρθρο 3 του πρωτοκόλλου, συνημένου στην Σύμφωνια προσχώρηση, λέει ότι ενδέχεται να έχει κάποιε ευθύνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εγώ ω μέλο του ελεγκτικού συνεδρίου δεν μπορώ να το σχολιάσω το θέμα, αλλά υπάρχει μάλλον ένα θέμα εδώ. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ανάγκη στην Λιθουανία να λάβει μέρο τη ευθύνη και η Κομισιόν, αυτό εξαρτάται όμω από την ερμηνεία του πρωτοκόλλου. Πάντως στην σύσταση 5 είμαστε σαφείς και κύριε Φόξ έρχομαι στο δεύτερο ερώτημά σας για το οποίο θέλω να πω δύο πράγματα. Ε, είναι το ερώτημα κατά πόσον αξιοποιήθηκαν σωστά τα χρήματα των φορολογουμένων. Το λέμε νομίζω σαφώς στην σύσταση 5. Πολλές φορές προτείνουμε ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός να σταματήσει. Και αυτό λέμε και στο 5. Διότι δηλαδή δεν πιστεύουμε ότι έχει αποτελέσει το κατάλληλο κίνητρο. Ίσα ίσα οδηγηθήκαμε σε καθυστερήσεις, επικαθυστερήσεων και μάλιστα προέκυψε και ένα μεγάλο χρηματοδοτικό κενό στην Λιθουανία. Οπότε, εκεί καθίστερε σαφές ότι δεν πιστεύουμε ότι ο σημερινός χρηματοδοτικός μηχανισμός έχει παράσχει τα απαραίτητα κίνητρα, θέλετε. Οπότε προτείνουμε να καταργηθεί. Κύριε Κόλτσεκ, πώς συγκρίνεται ο παροπλισμός στη Γερμανία, είπατε, με τον παροπλισμό στη Βουλγαρία ή σε χώρες με πρώην Σοβιετικούς αντιδραστήρες. Κοιτάξτε, εμεί δεν ελέγξαμε τη διαδικασία στην Γερμανία, τη διαδικασία παροπλισμού. Οπότε αυτά που θα πω είναι κάποια προσωπικά σχόλια και η Κομισιόν θα σχολιάσει ενδεχομένω και αυτή. Η μόνη αντιδραστήρες που παροπλήσαμε τώρα είναι η γερμανική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστος ήταν ε, λίγο πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανά αντιδραστήρα. Ανά αντιδραστήρα. Θα λέω ότι το πόσο που θα χρειαστούμε για του Σοβιετικού αντιδραστήρε δεν θα είναι μεγαλύτερο. Όμω οι γερμανικοί αντιδραστήρε είναι διαφορετικοί από αυτού του παλιού Σοβιετικού. Θα είναι λοιπόν ε, πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε ένα μοναδιαίο κόστος, ακόμη και αν είχαμε κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς. Πάντως, ε, οι πιο πεπειραμένοι στον τομέα αυτό στην Ευρώπη είναι οι Γερμανοί. Αυτοί έχουν ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο από την αρχή ως το τέλος, οπότε αυτό παίρνουμε και ως μπούσουλα στο μέλλον. Κύριε Μποσέκ, με ρωτήσατε σχετικά με την κλίμακα των παραπλησμών σε άλλες χώρες της Ευρώπης και αν υπάρχει δυνατότητα οικονομιών κλίμακας. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Στην σελίδα 17 συγκεκριμένα λέμε ότι είτε το θέλουμε είτε όχι. Η αγορά αυτή μεγαλώνει. Σε τέλη του 15, υπήρχαν 129 δραστήρες στην Ευρώπη και άλλοι 91 που είχαν κλείσει. Μάλιστα τρει είχαν παροπληστεί ήδη και 50 από τους 129 που είναι λειτουργία θα φτάσουν στο τέλο της ωφέλιμης ζωή του ως το 2025. Πολλοί θεωρούν ότι ο προπολισμός ενό συνδεδεστήρα δεν είναι οικονομική ανάπτυξη, αλλά κοιτάξτε, το ίδιο τελικά είναι. Όπω κατασκευάζει κανεί έναν αντιδραστήρα, έτσι τον αποσαρμολογεί, τον παροπλίζει. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο απασχολεί πολλού εργαζομένου. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα είναι να δει τον τομέα του παροπλισμού πυρηνικών αντιδραστήρων ω ένα τομέα οικονομική δραστηριότητα, όπου υπάρχει δουλειά. Να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτέ τι ευκαιρίε, ευκαιρίε μεταξύ άλλων απασχόληση. Οπότε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά για την ερώτηση αυτή. Ζήτησατε και μία διευκρίνηση όσον αφορά κίνητρα, γιατί έλεγα ότι ο παρόν χρηματοδοτικό μηχανισμό δεν παρέχει αρκετά κίνητρα κλπ. Μπορεί ορισμένοι από εσά να γνωρίζετε το γεγονό ότι μέρο τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι στο πλαίσιο συγχρηματοδοτημένων προγραμμάτων, όπω γίνεται στα ε, διαφορετικά προγράμματα. Τι εννοώ λοιπόν κίνητρα. Αν δώσετε λεφτά <laughs> δωρεάν οι άνθρωποι συμπεριφέρονται διαφορετικά σε σύγκριση με την κατάσταση όπου οι άνθρωποι βάζουν και δικά τους χρήματα. Τους νοιάζει περισσότερο. Γιατί αυτός που βάζει και αυτός δηλαδή χρήματα σε ένα έργο θα φροντίσει το έργο αυτό να ολοκληρωθεί. Ε, υπάρχει μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με τα δωρεάν χρήματα που ρέουν χωρίς κόστος δηλαδή. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Και για την ασφάλεια πριν και μετά τη Φουκουσίμα. Έχετε δίκιο ότι η σύμφωνη προσχώρηση υπεγράφει πριν από τη Φουκουσίμα. Εννοείται. Όμω, αν δεν κάνω λάθο, και τότε ήδη είχε γίνει μια συζήτηση σχετικά με το αν έπρεπε να κλείσουν αυτοί οι αντιδραστήρε, αλλά αυτό αποτελεί πλέον παρελθόν. Το θέμα είναι ότι από τι υποσημειώσει περάσουμε στην σκληρή πραγματικότητα ότι οι πρώην αυτοί οι σοβιτικοί αντιδραστήρε δεν πληρούν τι προδιαγραφέ ασφαλεία. Τώρα, ανεξαρτήτω το αν είναι πριν ή μετά τη Φουκουσίμα, όλοι κλείνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω. Και τέλο, ένα σχόλιο επί τη ερωτήσεω του κυρίου Χέγγελ όσον αφορά αυτό που σχολήσει και η Κομισιόν. Κοιτάξτε, θέσαμε το ερώτημα ω ελεγκτέ, γιατί μα απασχολεί το μέγεθος του έργου και δώσει μακροπρόθεσμη αποθήκευση. Εδώ τώρα ακόμα είμαστε στην αρχή φυσικά, στο στάδιο του σχεδιασμού. Όπως όμως είπατε και εσείς και συμφωνώ, δεν έχει νόημα όλα τα κρατημέλη να κάνουν το ίδιο πράγμα ξεχωριστά. Ε, όλε οι φορέ εμπλέκονται, γιατί υπάρχουν και τα ρευδιαργά ισότοπα, στα νοσοκομεία κλπ. Αλλά φυσικά έχουμε κυρίω τι χώρε που διαθέτουν πυρηνικού αντιδραστήρε. Έλεγα λοιπόν ότι δεν έχει αναγκαστικά νόημα κάθε χώρα να σκάψει μια τρύπα στο, στη χώρα της και να θα ψυχεί τα απόβλητα. Γιατί σε πολλές χώρες δεν υπάρχουν, δεν συντρέχουν και οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Προσωπικώς λοιπόν θεωρώ ότι είναι λογικό να κάνουμε κάτι σαν αυτό το οποίο έκανε η Κομισιόν και το οποίο περιγράφει σε ένα έγγραφο πριν από δύο εβδομάδε. Δηλαδή να δρομολογήσουμε έναν διάλογο με τα κράτη-μέλη για να διερευνήσουμε ε, κατά πόσο κάποιε περιφερειακέ λύσει είναι πλέον ενδεδειγμένε. Και το πράξαμε αυτό στο πλαίσιο τη εσωτερική αγορά ενέργεια, επί τη οποία ε, έχω μιλήσει στο παρελθόν στην Επιτροπή σα. Διερευνούμε και προτείνουμε περιφερειακές λύσεις και για λόγους ε, ενεργειακής ασφάλειας. Εκεί πετύχαμε και πιστεύω ότι γι' αυτόν τον λόγο πρέπει η ίδια αρχή να πριτανεύσει και εδώ για να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Αυτά ελπίζω να πίνετε σε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όμαν που ήρθατε καταρχήν και που καταθέσατε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις. Κύριος Κοχλιτσέκ, παρακαλώ. Μια παρατήρηση. Νομίζω κάνετε λάθος. Λόγω των αντιδραστήρων, των γερμανικών αντιδραστήρων, αναφέρεται ότι και οι σοβιετικοί αντιδραστήρες λειτουργούν, μάλλον ψύχονται με νερό σε στήλες και το θέμα είναι τι προστασία εξασφαλίζουμε με αυτήν την μέθοδο. Έχουμε ράβδου περιβαλλομένε από νερό. Αυτές οι ράβδοι μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα υπόλοιπα όμως είναι ραδινεργά απόβλητα. Δηλαδή, θέλω να πω, αν συγκρίνεται αυτούς τους απερχιωμένου αντιδραστήρες που ψήφονταν ε, με νερό κλπ. Ε, αυτοί οι δραστήρε έχουν το ίδιο πρόβλημα. Τεράστιε ποσότητε αποβλήτων που κάπου πρέπει να αναποτεθούν. Γι' αυτό και ρώτησα προηγουμένω. Και νομίζω δεν απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ και ευστό μα. Συγγνώμη που άργησα. Αλλά εδώ έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα που χρονολογείται από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Έχουμε ευκαιρία απασχόλησης, αλλά ποιος έχει βάλει στην άκρη και τα χρήματα για να πληρώσει το έργο. Έχουμε μεν μια εσωτερική αγορά, όπου Κανείς ε, αυτή την εποχή εγκαθιστά φωτοβολταϊκά ή ολικά πάρκα κλπ. Χωρίς σκέφτεται το, το μέλλον. Θέλω να πω ε, και σε αυτού του τομεί, τα φωτοβολταϊκά και αλλού, κανεί δεν βάζει λεφτά αυτή τη στιγμή στην άκρη για την ανακύκλωση όταν θα χρειαστεί. Ενώ βάζουμε λεφτά για την ανακύκλωση των τηλεοράσεων. Λοιπόν, στην δεύτερη οδηγία, στην οποία ήμουν εισηγητή, είχε προταθεί ένα τέτοιο ταμείο όταν, για όταν φτάσουν αυτές οι εγκαταστάσεις στο τέλος της ωφελημής ζωής τους. Εγώ ανησυχούσα ότι δεν έχουμε χρήματα. Και η Κομισιόν την εποχή εκείνη δημοσίευσε γραπτή δήλωση με την οποία ήταν κατά του μέτρου αυτού. Μας υποσχόταν όμως νομοθετική ρυθμίση κάποια στιγμή να λυθεί το θέμα. Και όμως 15 χρόνια αργότερα αυτή είναι η απάντησή του και, ή η εντυπωση μου και δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι από αυτό. Ε, εδώ έχουμε ένα κενό δισεκατομμυρίων, τριψήφιο θεωρώ. Λοιπόν, αν δεν πληρώσει κάποιο, ποιο θα πληρώσει οι καταναλωτέ πάλι. Είναι πρόβλημα τη εσωτερική αγορά και τη Κομισιόν. Και η Κομισιόν, επαναλαμβάνω, δεν, δεν έκανε ποτέ τίποτα σχετικά με το θέμα. Ευχαριστούμε. Οπότε να δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο να δώσει τις ε, τελευταίες απαντήσεις <clears throat> σε αυτά τα τελευταία ερώτημα. Καταρχήν ε, να ζητήσω συγγνώμη από τον κύριο Καλέτσακ. Ε, πράγματι είχατε και Θα έπρεπε να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν προ... σε έλεγχο των γερμανικών καταστάσεων. Με διορθώσατε σε σχέση με αυτό. Πράγματι ο έλεγχος που κάνατε εσείς ήταν καλύτερος από το δικό μας, οπότε σας ζητώ συγγνώμη. Τώρα σε ό,τι αφορά αυτούς τους αντιδραστήρες. Ουσιαστικά δηλαδή αυτοί που είναι στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία, που βρίσκονται στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία, είναι παρόμοιοι με αυτέ του Σοβιετικού τύπου που αναφέρατε, αλλά εκείνος, εκείνη στη Λιθουανία δεν είναι. Ε, και βλέπω πω ε, συνεννείται. Καλώ. Ε, σα ευχαριστώ για αυτή τη διόρθωση σε ό,τι αφορά ακριβώ την διαφορά και με του αντιδραστήρες τη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ερώτημα θα δώσουμε και το λόγο στην Επιτροπή. Πρώτο από την πλευρά του ελεκτικού συνεδρίου ε, ε, να σας ε, παραπέμψω στη στήσταση 8, όπου λέμε ότι θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια και σαφήνεια ως προς το ποιος φέρει την ευθύνη, έτσι ώστε και εμείς ως ελεγκτής να γνωρίζουμε ότι υπό την ευθύνη κάποιου εκτελείται ένα έργο, γιατί εκεί βρίσκεται ακριβώς η απαρχή της επίλυσης ενός προβλήματος. Ακριβώς λοιπόν αυτό αναφέρουμε στην έκθεση, ότι ορισμένες φορές δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν ο υπεύθυνο φορέας για τις διαδικασίες. Επιτρέψτε όμως να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέω ο Πρόεδρος. Ο κύριος ε, Γεράσιμος Θωμάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κύριο Τόμας για αυτό το ερώτημα. Ναι, νομίζω πως η κατάσταση έχει βελτιωθεί από εκείνο το στοίχημα που ανέφερα εδώ Ευρωβουλευτή. Ε, την τελευταία εβδομάδα υποβάλαμε στο Κοινοβούλιο την έκθεση ό,τι αφορά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την εκτέλεση τη οδηγία για τα πυρηνικά, είπαμε τώρα διενεργά απόπλητα και είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται αυτή η έκθεση. Οπότε νομίζω πω θα πρέπει να αποτελέσει ε, αντικείμενο περαιτέρω συζήτηση. Όμω αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση ότι με βάση τι πληροφορίε που έχουμε λάβει από όλα τα κράτη-μέλη, το κόστο εκτιμάται ε, σήμερα ημέρα στα 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε συλλέξει τις πληροφορίες, τα δεδομένα από όλα τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τα απόβλητα και το κόστος της διαχείρισης ε, των αναλωμένων καυσίμων και των αποβλήτων. Δυστυχώς, στο πλαίσιο της ε, διαβούλευσης που έγινε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, δεν έγινε δεκτή η πρόταση που είχε κάνει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εναρμονισμένη υποβολή εκθέσεων. Οπότε χρειάστηκε εμεί να κάνουμε κάποιου υπολογισμού από μόνοι μα ω Επιτροπή. Πάντω, εδώ έχουμε τι πρώτε εκτιμήσει σε ό,τι αφορά το κόστο, ε, ποια είναι τα. Ε, τα μία, δηλαδή τα κονδύλια τα οποία έχουν συγκεντρωθεί προς αυτό το σκοπό και τα οποία δεν επαρκούν και αναφέρουμε επίσης ότι ακριβώς θα χρειαστούν συμπληρωματικές δράσεις, προγράμματα από την πλευρά των κρατών μελών για να ε, πληρωθεί αυτό το χάσμα. Και σε τρία έτη θα επανέλθουμε ε, με μια νέα έκθεση όπου θα αναφερόμαστε στους τρόπους αντιμετώπισης ε, αυτού ακριβώς του χρηματοδοτικού χάσματος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Διευθυντή και ευχαριστούμε τον κύριο Γουλόου εδώ για την παρουσίαση που μας έκανε και τις απαντήσεις που μας έδωσε που ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και βέβαια και πολύ σημαντικές για την ασφάλειά μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ότι καλύτερο. Περνάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διαταξής μας η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, που αποτελεί τμήμα του χειμερινού πακέτου, όπως λέγεται, ή του ε, πακέτου της καθαρής ενέργειας για όλους. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και επιτρέψτε μου να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σχέδιο εκθεσής σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ε, εισηγητής ο κύριος Μπέντσεν και πρόκειται για την ε, πρώτη έκθεση που έχει ως αντικείμενο ακριβώς αυτό το πακέτο καθαρής ενέργειας για όλους, που αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από την πλευρά της Επιτροπής Ήτρε. Δίνω το λόγο λοιπόν στον συνάδελφο Κρικ Μπέντσε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και ευχαριστώ τους σκιώδει συγητές, την Επιτροπή και όλου του ε, συναρμόδιου εφορείς ε, που συνέβαλαν στην διαδικασία σύνταξης αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους σκιώδει συγητές που από νωρί συμμετείχαν στη σύνταξη του σχεδίου έκθεσης. Ε, ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι ότι τα κτίρια συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εσωτερικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση αλλά και την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών. Αυτή λοιπόν η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ε, έχει ένα σημαντικό δυναμικό σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, τη μείωση των ενεργειακών εισαγωγών ε, από την Ευρώπη, ε, χαμηλότερα τιμολόγια χρήσης ενέργειας ε, για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο υγιείς και αποδοτικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, αλλά και δημιουργία θέσεων εργασίας και υποστήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Τα κύρια στοιχεία λοιπόν εδώ του σχεδίου έκθεσης εστιάζουν σε, τρεις, σε τρία θεματικά πεδία. Πρώτον, εξασφάλιση υψηλότερη δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών με συγκεκριμένε απαιτήσει σε ό,τι αφορά την κινητικότητα με ηλεκτροκίνητα οχήματα και ε, την παροχή των καταλλήλων κινήτρων για αναγεννήσει. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ε, θεματικό πεδίο, ε, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις των κρατών μελών, αναφέρουμε ότι ο στόχο του MPD θα πρέπει να είναι κατασκευή κτηρίων που είναι εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτικά και με χαμηλέ ανθρακούχε εκπομπέ. Εδώ ε, προτείνουμε να υπάρξουν και κατάλληλε εθνικέ στρατηγικέ με, ε, με τον απαιτούμενο σεβασμό της διαφορετικότητας ε, της ενέργειας ε, στην Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη και την αλληλεγγύη. Επίσης προτείνουμε να λάβει υπόψη η ενεργειακή ένδυα ε, και η κατανομή περαιτέρω κινήτρων καθώς και η αύξηση των σχετικών δεξιοτήτων και η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ελόγω αγορά. Χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια που θα εισρέψουν σε αυτή την αγορά. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν το πώς οι δικές τους στρατηγικές ανακαίνισεις θα συμβάλλουν στους στόχους ενεργειακής απόδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρξει και η κατάλληλη αποτελεσματική περικοπή των δαπανών τους. Τώρα, στο δεύτερο θεματικό πεδίο σε ό,τι αφορά δηλαδή, την ε, κινητικότητα με ηλεκτροκίνητα οχήματα, νομίζω πως είναι μεγάλη ε, φιλοδοξία εδώ όλος μας να υπάρξει ακριβώς περισσότερη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στα μέσα μεταφορά ε, για να μειώσουμε τις ανθρακούχε εκπομπές. Ε, τα όσα μας προτείνει η Επιτροπή σε ό,τι αφορά την κινητικότητα και τη σχετική υποδομή δημιουργούν ανησυχίε σε ό,τι αφορά δηλαδή ε, το ποιοι θα είναι οι συναρμόδιοι φορεί, πώς θα γίνει η περικοπή των εσόδων, πώ θα παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα. Γι' αυτό λοιπόν προτίζουμε στην έκθεσή μα να υπάρξει σχέση με τις κατάλληλες ε, καινοτομίες αυτής της χρηματοδότησης και της υποστήριξης έτσι ώστε να μην υπονομεύσουμε τις ε, προσπάθειες ε, καινοτομίες. Επίσης, Επίσης προτείνουμε να υπάρξει και περισσότερη υποστήριξη του free tube ώστε να υπάρξει ε, περαιτέρω ε, συμπίεση των δαπανών και να μην υπάρχει δηλαδή μόνο και μόνο χρήση των σταθμών ε, ανεφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τρίτο στοιχείο, το τρίτο που αναφέρουμε στο σχέδιο έκθεση, είναι το εξή. Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι υπάρχει ανησυχία ότι τέτοιου είδου καινοτομίε είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο απευθύνεται μόνο στου ε, πλουσίου ε, και του προνομιούχου. Εμεί αντιθέτω, όταν κάνουμε λόγο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, δεν κάνουμε λόγο μόνο για την ε, μόνωση κτηρίων ή τη χρήση, για παράδειγμα, υψηλών τεχνολογιών σε κτίρια. Θεωρούμε, και φρονώ εγώ ίδιο, ότι υπάρχουν μία σειρά από τροποποιήσει προσιτές σε κόστος που μπορούν να διεξαχθούν από τους ιδιοκτήτες κάποιων ακινήτων ε, που ξεκινούν από, το 20, από τα 20 ευρώ για να δώσω ένα παράδειγμα. Οπότε για να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι ώστε να υπάρξει δηλαδή ανακαίνιση, ε, ενεργειακή ανακαίνιση σε μικρά, σε, μικρές, σε μικρά και μεγάλα κτίρια. Οπότε θα πρέπει να αποφύγουμε ε, διαδικασίες οι οποίες θα είναι αντιπαραγωγικές σε ό,τι αφορά την παροχή σχετικών κινήτρων. Και τι εννοώ εδώ, ε, εδώ υπερβολικές απαιτήσει, ε, ελλειπής διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει επιθεώρησης και ε, κατάλληλοι υπολογισμοί σε ό,τι αφορά το σύνολο της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Κλείνοντας, Πρόεδρε, να πω ότι αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία που θα έχω με τους κοιόδους ηγητές, τους υπολείπους συναδέλφους, την Επιτροπή και του ε, συναρμόδιου φορεί και χαιρετίζω τη συζήτηση που θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά τις ε, ε, τροπολογίε που θα υποβληθούν πριν ή έω την προθεσμία υποβολή του, δηλαδή στις 8 Ιουνίου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος θα είναι μικροφώνου. Ευχαριστώ. Εγώ με χαρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή ο οποίος ήταν πολύ προοδευτικό σε ό,τι αφορά τη σύνταξη τη έκθεση, αλλά και το γεγονό ότι ήταν διατεθειμένος να συνεργαστεί από νωρί ε, με του σκιώδεις εισηγητές. Ε, πραγματικά το επιχειρώ αυτό. Ε, έκανε μια αναφορά στην ενεργειακή ένδυα, ε, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για τη δική μα πολιτική ομάδα και θα ήθελα να το αναφέρω πρώτο. Δηλαδή είναι, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σύνολο αυτή τη έκθεση, η ενεργειακή ένδυα και γίνεται μια συγκεκριμένη πρόταση όπου όταν δηλαδή θα, το κάθε κράτος μέλος ε, θα συντάσει την στρατηγική του, εθνική στρατηγική για την ανακαινήση, πρέπει να λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη του ε, τα ε, κτίρια με τη χειρότερη ε, απόδοση. Οπότε εδώ θα θέλαμε να τροποποιηθεί περαιτέρω το σχέδιο έκθεση, ώστε να κάνουμε καλύτερη, ε, πιο εμφατική αναφορά στην ενεργειακή ένδυα. Μια ένδυα, η οποία βέβαια ε, κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, αλλά παραμένει σημαντική για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ταχύτητα τη κατασκευή νέων εκτηρίων, να πούμε ότι οι ρυθμοί είναι ακόμα βραδύ. Οπότε ο στόχο εδώ του εισηγητή είναι να επιταχυνθούν αυτοί οι ρυθμοί. Γιατί βέβαια γνωρίζουμε ότι το 40% τη ε, Χρήση τη ενέργεια ακριβώ απορροφάται από τα κτίρια και το 30% από τι μεταφορέ, οπότε θα πρέπει πάντοτε να αναφέρουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να υποστηρίξουμε τι σχετικέ δράσεις. Για παράδειγμα, για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα χρειαζόμαστε και την κατάλληλη υποδομή. Και την υποδομή εκείνη η οποία θα είναι πιο αποδοτική και από άποψη ε, κόστου. Θα έχει την καλύτερη σχέση κόστου αποτελέσματο. Η ε, πρόταση δηλαδή τη Επιτροπή είναι υπερβολική αρκετά φιλόδοξο όταν μας λέω στο 2025 ότι δηλαδή θα πρέπει να, υπάρχουν, ε, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη υποδομή δηλαδή για, ε, για τα ηλεκτρικά οχήματα παντού. Εντάξει, είναι φιλόδοξη από τη μία πλευρά αυτή η πρόταση της Επιτροπής, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε τα όσα προτείνονται. αλλά βέβαια ε, κανείς αγοράζει ένα αυτοκίνητο όχημα μόνο εφόσον υπάρχει και η κατάλληλη υποδομή και το αντίθετο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει υποδομή δεν αγοράζει κανείς ένα τέτοιο όχημα. Όμως, από εκεί και μετά, παρότι το, οι δράσεις είναι θετικές, θα ήθελα να υπάρχει, ε, να διασφαλιστεί συνοχή μεταξύ των επιμέρους ε, δράσεων ε, και να υπάρχει και το μεγαλύτερο όφελος για τους καταναλωτές. Θεωρούμε πως συχνά η κατοχή των κτηρίων που δεν είναι δεν κατοικούνται δηλαδή, είναι, είναι επαγγελματική ε, χρήση, ε, ε, βρίσκονται στα χέρια, οι κατοχήνε επιχειρήσει. Οπότε εκεί θα πρέπει να. ενδεχομένως να προβλέψουμε ψηλότερε απαιτήσει γιατί εκεί ακριβώς είναι εύκολο να αποσβεστούν τα σχετικά, οι σχετικές Επίσης σε ό,τι αφορά την υγιή ποιότητα αέρα και την αναφορά που είχε γίνει σχετική έκθεση της ΣΥΤΡΕ να πούμε ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, αξιώνοντα από τη μία πλευρά υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των ιστορικών των κτηρίων και από την άλλη υψηλότερη, για παράδειγμα, παρουσία μούχλα λόγω εργασία στα κτίρια. Από εκεί και μετά θα ήθελα να προτείνω μια τροπολογία έτσι και απο τροφή για σκέψη. Ενδεχομένως δηλαδή εδώ η Ήτρε να συνδυάσει τι εργασίες που κάνει από τη μία πλευρά για την ενέργεια και από την άλλη πλευρά για την ψηφιακή μετάβαση, ε, digital transform. Οπότε εγώ, εγώ, εδώ έχουμε και έναν ε, δείκτη της αγοράς, τον οποίο αναλύει ο εισηγητής, αλλά πέραν αυτού ενδεχομένω θα μπορούσαμε να περιλάβουμε κάτι. Για παράδειγμα, δηλαδή υψηλή απόδοση συνδέσει ή για παράδειγμα συνδέσει μέσω οπτικών ινών, οι οποίε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο τη ανακαίνιση των κτηρίων για του σκοπού τη ενεργειακή απόδοση. Δηλαδή, όταν γίνεται μια τέτοια ανακαίνιση, γιατί ταυτόχρονα να μην υπάρχει και ένα προπολογισμό στο πόσο θα κόστιζε αυτό το κτίριο να ε, συνδεθεί και ψηφιακά μέσω ε, οπτικών νόμων. Πρόκειται δηλαδή για ένα στοιχείο το οποίο δεν βρίσκεται ε, αποκλειστικά στα πλαίσια της, αυτού του πακέτου για την ενεργειακή απόδοση, αλλά στα γενικό, στους γενικότερους στόχους που έχουμε uh, Ευχαριστώ κύριε από την Άλντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για μια πολύ καλή έκθεση που μας παρουσίασε, μισορροπημένη και χαίρομαι που δείτε πρώτα έμφαση στην ενεργειακή απόδοση. Και βλέπω ότι λαμβάνουμε υπόψη μας και άλλα στοιχεία εσωτερικά το κερίον δηλαδή. Αυτό είναι πρώτη φορά και νομίζω είναι πολύ καλό. Και νομίζω ότι είναι καλό επίσης να έχουμε τις οι πράξεις για την έκθεση αυτή από τη στιγμή που έχουμε μια έννοια αρκετά δυναμική και ενεξελίξη που ερμηνεύεται ενδεχομένω διαφορετικά στις χώρες μέλη. Επίσης νομίζω ότι είναι καλό να μετατοπίσουμε τις υποχρεώσεις στις χώρες μέλη και να τις υποχρεώσουμε να υποβάλουν τις δικές τους έτσι, σκέψεις, απόψεις και σχεδιασμό σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και τα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουν οι ίδιες χώρες μέλη τις δικές τους προθέσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Να αναφερθώ σύντομα σε δύο ζητήματα. Καταρχάς ΑΠΕ και να κάνω κάποια σχόλια για τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση για τις μηδενικές προδιαγραφές δηλαδή η παραγωγή επιτόπου από εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε σχέση με πιο ολιστική προσέγγιση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν εμείς επιμείνουμε σε συγκεκριμένους στόχους για την επιτόπου παραγωγή ΑΠΕ αντί για, αντί για μια πιο οριζόντια προσέγγιση τότε νομίζω υπονομεύουμε το βάρος των ΑΠΕ. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή αυτή τη σχεδόν ε, μηδενική πρωτογραφή σε σχέση με μια πιο ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση των ΑΠΕ στις κατοικίες. Μετά για τους πρωτογενείς παράγοντες ενέργειας και πάλι νομίζω ότι θα έπρεπε να βελτιστοποιήσουμε το μερίδιο των ΑΠΕ συνολικά και για τις κατοικίες. Κάτι το οποίο βεβαίως οδηγεί σε συζητήσεις τώρα για το κατά πόσο από τώρα θα πρέπει να δούμε τους πρωτογενείς παράγοντες ενέργειας στην έκθεση. Αυτό είναι κάτι θα πρέπει να το συζητήσουμε θέλω νομίζω Σάλτε. Και τέλος, δύο παρατηρήσεις για τη χρηματοδότηση. Νομίζω θα πρέπει να απελευθερώσουμε το δυναμικό που υπάρχει όσον αφορά τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων. Κάτι το οποίο πρέπει όμως να συνοδεύεται από μακροχρόνιους στόχους και διαβεβαιώσεις όσον αφορά την ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων ενεργειακή απόδοση για τι κατοικίε. Και θα πρέπει επίση να ενσωματώσουμε αυτό που κάνει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με το ΕΦΣΥ, ώστε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά με τα ενδεχόμενα ιδιωτικά κεφάλαια που θα ενδιαφερθούν. Αυτό θα θέλαμε να κάνουμε και να τα κάνουμε συνδυαστικά. Ξαναλέω λοιπόν, πολύ καλή έκθεση. Θα εξετάσουμε περαιτέρω και λεπτομερέστερα κάποια στοιχεία που αφορούν τις ΑΠΕ και τις κατοικίες και να δούμε περισσότερο επίσης και τα θέματα χρηματοδότηση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μας αλέσει, ε, ε, των Πρασίνων. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριο Μπέντσεν για την έκθεσή του. Επειδή ήταν πολύ περιεκτικός με όλες τις πολιτικές ομάδες και ιδιαίτερα με τους πράσινους και το ευχαριστώ για την διάφανη μεθοδολογία του σε σχέση με αυτό το θέμα. Εκ μέρους των πρασίνων να αναφερθώ συγκεκριμένα σε τρεις άξονες. Καταρχάς η ολιστική σφαιρική προσέγγιση, δεύτερον φιλοδοξία και τρίτον η ανθρώπινη διάσταση. Να ξεκινήσω πρώτα με τη φιλοδοξία. Επειδή θεωρούμε ότι μετά τη Συμφωνία του Παρισιού που επικυρώσαμε πριν από λίγο, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο φιλόδοξοι. Ο στόχος της έκθεσης θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 40% όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Επίσης, για την καινοτομία αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό το 40% θα πρέπει εδώ να περιλάβουμε όλες τις κατοικίες και τις κοινωνικές κατοικίες και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τη στρατηγική ανανέωσης μακροπρόθεσμα. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για μας, ώστε να έχουμε έτσι την κατάλληλη προσέγγιση εκ μέρους της Ένωσης μετά τη Συμφωνία του Παρισιού. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μεμονωμένα στις κατοικίες, στα κτίρια. Το κτίριο καταρχάς ανήκει στην συνοικία και στο αστικό περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να το ανακαινήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή απόδοση, αλλά απόδοση του συνόλου στο οποίο ανήκει ένα κτίριο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα διάφορα συστήματα ψήξη, θέρμανσης κλπ. Θα ήθελα επί τούτου να κάνω δύο προτάσεις. Καταρχά σε σχέση με το Near Zero Energy Building θα πρέπει να πούμε το ίδιο και στο ευρύτερο πλαίσιο δηλαδή στην συνοικία, όλη τη συνοικία στην οποία ανήκει ένα κτίριο. Μετά, μεταφορές. Για τις μεταφορές θα πρέπει μόνο να δούμε τι γίνεται με τις μεταφορές με ηλεκτρικά οχήματα, αλλά την βιώσιμη, τις βιώσιμες μεταφορές. Να δούμε τι γίνεται με τα άτομα, δημόσιες μεταφορές, μέσα μαζικών δηλαδή μεταφορών, ποδήλατα, η εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών ώστε να υπάρχει βιωσιμότητα. Και τέλος, η ανθρώπινη διάσταση. Μιλήσατε για την ενεργειακή φτώχεια, κάτι το οποίο μας φαίνεται θεμελιώδες και θα κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε αυτή ακριβώς την πτυχή που σχετίζεται και με την υγεία. Θα ενισχύσουμε επίσης και τα τμήματα που αφορούν την κατάρτιση των εργαζομένων στα κτίρια, στο εσωτερικό των κτίριων και αυτό είναι απαραίτητο και επίσης θα θέλαμε να θέσουμε στο επίκεντρο αυτής της ε, μεταρρύθμισης τους πολίτες. Αυτούς δηλαδή που θα κάνουν αυτή την ενεργειακή επανάσταση. Οπότε θα πρέπει να έχουμε δύο είδη φορέων τις ε, συνεταιριστικές οργανώσεις στην ενέργεια αφενός και τις πόλεις. Πόλεις που είναι οι φορείς της ενεργειακής επανάστασης από κάτω. Θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να ακολουθήσουμε τις κατευθυντές γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισότητα φύλου και στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα όσον αφορά το χειμώνα. Θα είχα και σχόλια, να κάνω σε σχέση με το διαβατήριο που ακούσαμε ως ε, πρόταση και άλλες προτάσεις, το ΠΕΦ και τους δείκτες που αναφέραμε. Αλλά να καταλήξω λέγοντας το εξής. Η τεχνολογία αυτή χαμηλή ένταση στο OTEC, είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για τα πιο ε, φτωχά σύνολα κατοικιών, αλλά για το σύνολο του πληθυσμού, ώστε να υπάρχει τεχνολογική προσαρμογή σε όλες τις κατοικίες και σε αυτό το θέμα θα επιμείνουμε στις τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστώ, Σάλφε. Ο κύριος ε, για το προσχέδιο της έκθεσης που κατάθεσε, αλλά να σημειώσω επίση την επικοδομητική συζήτηση που είχαμε στην πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών. Για την ομάδα μα αποτελεί η προτεραιότητα να επιταχυνθεί η ανακαίνιση για την ενεργειακή αποδοση των κτηρίων, ώστε έτσι να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει για την προστασία του περιβάλλοντο, αντιμετώπιση δηλαδή των κλιματικών αλλαγών, και ταυτόχρονα επιτύχουμε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση ε, για προστασία της υγείας των ανθρώπων που ζουν σε παλαιά κτίρια με βλαβερές κλιματικές συνθήκες. Για μας, για την ΚΟΕ, είναι σημαντικό ε, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης να συμβάλλει μέσω συγκεκριμένων μέτρων και στη μείωση του κόστους που καλούνται να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Ε, και κατ' επέκταση εννοείται στην καταπολέμηση της ενεργειακής στόχιας. Δεν πρέπει να ξεχάνουμε ποτέ ότι είναι ένα σημαντικό στόχο αυτού, δεδομένου ότι σήμερα 23 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ένωση ζουν σε συνθήκε ενεργειακή στόχη. Επίση, πρέπει να διασφαλίσουμε πω οι αλλαγέ που θα επέρθουν με την νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με προσιτό κόστο για του ιδιοκτήτε. Ιδιαίτερα οι ευάλωτε ομάδε θα πρέπει να στριχτούν οικονομικά ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στι απαραίτητε ανακαινήσει και ταυτόχρονα να προωθήσουμε για τέτοια κτίρια και τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια μέσω επιδοτήσεων. Τώρα έρχομαι στα προβλήματα. Ιδιαίτερα προβληματική κατά τη γνώμη μα είναι η πρωτοβουλία έξυπνη χρηματοδότηση για τα έξυπνα κτίρια. Επί τη ουσία θα χρησιμοποιεί εγγυήσει του δημοσίου για να μοχλεύει ιδιωτικέ επενδύσει καθώ θα περιορίζει το ρίσκο των ιδιωτών. Κατ' επέκταση δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση πως οι επενδύσεις θα γίνονται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αλλά θα, γίνεται, θα γίνονται αυτές οι επενδύσεις εκεί που θα επιλέγουν οι ιδιώτες επενδυτές. Εμείς τονίζουμε ξανά πως πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα η χρηματοδότηση των κτηρίων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το κτηρίο σε υποβαθμισμένες και απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και το κτηρίο στις οποίες στεγάζονται μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά το προσχέδιο τη έκθεση που κατάθεσε ο συγητή, χαιρετίζομαι τι προτάσει για βελτίωση τη υγιεινή και του κλιματισμού των εσωτερικών χώρων, τι προτροπέ για αφαίρεση του αμοιάντου καθώ και άλλων επιβλαβών νησιών την υπογράμμιση πω πρέπει να συμπληρωθούν συγκεκριμένε ενέργειε που να συμβάλλουν στο περιορισμό τη ενεργειακή στόχιας, καθώ και στην επισήμαση πω τα κράτη-μέλη πρέπει να καθορίσουν στοχευμένε δράσει με μετρήσιμα αποτελέσματα για του καταναλωτέ που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδυα. Ωστόσο, έχουμε διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την πρόταση για τον δίχτυ ευφυία ω προτεραιότητα τη οδηγία. Επίση, δεν συμφωνώ πω τα μέτρα οικονομική βοήθεια πρέπει να εξαρτούνται από τα αποτελέσματα τη αναγέννηση. Αντιθέτω, όταν τα νοικοκυριά προχωρούν στι απαραίτητε ανακαινήσει, θα πρέπει να παίρνουν και τι προβλεπόμενε επιδοτήσει. Τέλο, δεν θεωρούμε πω πρέπει να τεθεί ω προτεραιότητα η δημιουργία υποδομών για επαναφόρτωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η πρόταση αυτή πρέπει να είναι προαιρετική, γιατί νομίζω για όλους μας είναι ξεκάθαρο ότι μια τέτοια, ε, ε υποδομές θα επιβαρύνουν με αχρίαστο, δυσβάσταχτο κόστος πολλά νοικοκυριά. Και πρέπει να πω, Πρόεδρο, ότι προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και οι τροπολογίες που θα καταθέσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you ε, Ευχαριστώ πολύ. Πλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ τα δικά μου συγχαρητήρια προς τον εισηγητή για την έκθεσή του. Όπως αναφέρει, η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό για τη μείωση της κατανάλωσης, βελτίωση της ασφάλειας και υποχώρηση των εισαγωγών ενέργειας και με τρόπο κερδοφόρο. Η έμφαση στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και οι δείκτες ευφυΐας νομίζω ότι είναι βελτιώσεις που ενισχύουν το κείμενο. Όμως, ως εισηγητής της έκθεσης για τις ΑΠΕ, απαραίτητο την ενίσχυση της υποδομής για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι βασικό για την απομάκρυση από τον άνθρακα και την πρόθεση των απέστης μεταφορές. Θα ήθελα επίσης να ακούσω λεπτομερέστερα δύο πράγματα για την 56 τροπολογία όσον αφορά τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο δίκτυο παραγωγής ενέργειας. Επίσης, να πω ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να απελάβουμε εδώ το θέμα της ενεργειακής στόχιας, θέμα πολύ σημαντικό και όπως είπε ο σοσιαλιστής συνάδελφος προηγουμένως θα πρέπει να ενισχύσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον συνάδελφο για το σχέδιο εκθεσής του για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Νομίζω ότι υπάρχουν ε, περιθώρια βελτίωσης στα νέα κτίρια και στα κτίρια στα προάστια. Θα πρέπει να δούμε επίσης τι γίνεται και με τα πάρκινγκ κατά διάρκεια των εργασιών που θα πρέπει να γίνονται. Εργασίες οι οποίες βέβαια όσον αφορά τα ηλεκτρικά κυκλώματα θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο τρόπο και εδώ ακριβώς ε, συμμερίζουμε και τις απόψεις του εισηγητή για τις τροπολογίες 29 και 30. Θα πρέπει επίσης να προσέξουμε για το θέμα της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό των νεοκτηρίων και θα πρέπει να ενισχύσουμε τις εγκαταστάσεις και το εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει το σωστό αερισμό των κτηρίων. Έχουμε επίσης και τους δείκτε ευφυΐας, οι οποίοι, οι οποίοι δεν θα πρέπει βεβαίω να επιφέρουν περαιτέρω κόστο για τους ιδιοκτήτε και θα πρέπει να αναπτύξουμε ευφυεί συστήματα σε κτίρια που δεν είναι κτίρια κατοικίας. Νομίζω ότι τα περιθώρια κέρδους είναι ενθαρρυντικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δανίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να διαβεβαιώσω τον εισηγητή ότι θα έχει την πλήρη υποστήριξή μας και να αναφερθώ σε κάποια κύρια σημεία για μας. Η ενεργειακή φτώχεια, καταρχάς. Θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό το θέμα. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το σημαντικό πρόγραμμα που έχουμε θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε και επίσης μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αποφύγουμε το να ανταποκρίνουμε στην ανάγκη αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη για περισσότερη βοήθεια. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε κάτι και για τα ηλεκτρικά οχήματα. Νομίζω δεν κάνουμε αρκετά πράγματα για αυτό το θέμα. Δεν είμαστε αρκετά τολμηροί. Ίσως στο μέλλον να εξελιχθούν τόσο γρήγορα τα πράγματα που θα έχουμε μείνει πίσω εμεί. και να βρεθούμε σε κακή κατάσταση. Γιατί αυτοί που θα αγοράσουν τα ηλεκτρικά, θα αγοράσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία θα έχουν ε, χαμηλότερε τιμέ, θα βρεθούν χωρί το απαραίτητο αριθμό σημείων φόρτιση. Αυτό θα πρέπει λοιπόν να το, το ρυθμίσουμε από τώρα. Θα πρέπει να το συνδέσουμε επίση και με το θέμα των νέων των κτηρίων, τα κτίρια που κτίζονται αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συνοδεύονται από σημεία φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια τάση η οποία εξελίσσεται και προχωράει συνέχεια. Οπότε εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα τη ε, οικονομικής ενίσχυσης στη Ρουμανία, α πούμε. Υπάρχει ένα ποσό επιδότηση 10.000 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το 2025 θα έχουν φτηνίνει τόσο οι τιμέ αυτών αυτοκινήτων που θα είναι φτηνότερα από τα κανονικά αυτοκίνητα. Αλλά δεν υπάρχουν σημεία φόρτιση. Πρέπει λοιπόν να ομονοούμε και με την Κομισιόν Γενική Διεύθυνση Ενεργική Ρέτζιο, οι οποίες δεν έχουν ακριβώς γνώση του τι κάνουμε εμείς εδώ. Στη Ρουμανία, να σα ξαναπώ, είχαμε ένα πρόγραμμα όπου βοηθήσαμε τη δημιουργία νέων κατοικιών που θα προβλέπουν την ύπαρξη αυτών των σημείων. 100.000 μάλιστα. Και νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο εδώ, αλλά βλέπουμε ότι η γραφειοκρατία είναι τεράστια σε αυτά τα προγράμματα της Ένωσης. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνουμε ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, χωρίς να έχουμε γραφειοκρατία να μας αποτρέπει να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στους ΟΤΑ πούμε, να διαχειριστούν όλο αυτό το θέμα γιατί νομίζω ότι είναι η να το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πρακτικές παρατηρήσεις. Το σχέδιο έκθεσης είναι πολύ ενδιαφέρον όμως αντιμετωπίζει το θέμα μάλλον θα έλεγα αφιψηλού δηλαδή πολλοί όπως είπε ο Σάδεφος Νίκας αξιοποιούν διάφορα προγράμματα ας φανταστούμε μεγάλο αριθμό διαμερισμάτων ιδιοκτήτων διαμερισμάτων εκεί ήταν πολύ δύσκολο να συμφωνήσουν όλοι οι διοκτήτε για μια τέτοια εγκατάσταση. Η διαπραγμάτευση, αν θέλετε, είναι σύντομα δύνατη. Πρακτικά, λοιπόν, στα σημερινά κτίρια. Τι συμβαίνει. Έχουμε εγκατεστημένη συνδεσμολογία, η οποία μπορεί να καταλήγει στην απαραίτητη πρίζα, στο σημείο φόρτισης αν θέλετε, στο ρευματοδότη. Εκεί μπορεί κάποιο που έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο να φορτίσει αργά αργά τη μπαταρία του. Βεβαίως, ε, αν θέλει κανείς ταχεία φόρτιση, αυτό προϋποθέτει παροχή 64 αμπέρ οποίο σημαίνει ότι χρειάζεται διαφορετική καλωδίωση. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι 32 ή 64 αμπέρ. Θα χρειαστούμε νέα καλωδίωση ή όχι. Τώρα για τους σκοπούς της ε, κινητικότητας. Καλό θα ήταν για να διευρύνουμε τον πληθυσμό των ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων, δηλαδή να περιοριστούμε στα 32 αμπέρ, με πηγή όμως τα φωτοβολταϊκά ή την ολική ενέργεια. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και η πηγή δηλαδή της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι μια φιλική προς το περιβάλλον. Αν η πηγή είναι ανανεώσιμη, σε αυτή την περίπτωση θα είναι λογικό να περιοριστούμε στα 32 αμπέρ για αυτοκίνητα των 30 κιλοβάτ περίπου. Από εκεί πέρα προς την ε, φτώχεια. Στα νέα κτίρια τα ενίκια είναι μάλλον υψηλά. Δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλοι. Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια ακριβή υπόθεση. Ύστερα Στις χώρες μας σχεδόν όλα τα νοικογύρια έχουν μια παροχή τουλάχιστον 6 αμπέρ. Το θέμα είναι θέλουμε τα κρατη να εφαρμόσουν μέτρα προς την σωστή κατεύθυνση ή όχι. Θα οθήσουμε τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση ή όχι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπένσον για την εξαιρετική έκθεση. Η δική μου αίσθηση είναι ότι στα νέα κτίρια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος. Ε, πολλά κτίρια είναι μηδενικών εκπομπών. Το θέμα είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό με τρόπο αποδοτικό. Το πρόβλημα είναι όμως τα υφιστάμενα κτίρια, τα παλιά κτίρια, όχι τα νέα. Και δεν είναι το πρόβλημα μόνο της Ρουμανίας. 80% των κτηρίων που θα υπάρχουν γύρω μας το 2050 υπάρχουν ήδη σήμερα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι κάνουμε για την ανακαίνιση αυτών των κτηρίων. Και δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει νέα λύση. Έχουμε διαφορετικά κτίρια σε διαφορετικές χώρες. Η λύση πρέπει να εξαρτάται από τη χώρα, από τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος είναι να εφαρμόσουμε χάρτες πορείας, για τα κτίρια για τα επόμενα χρόνια. Στην ε, προηγούμενη έκθεση η λύση που προτείναμε δεν ήταν 100% σωστή. Εν πάση περιπτώσει κάναμε μια καλή αρχή. Τώρα αν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι το σχετικό άρθρο δεν το εφάρμοσαν όλα τα κρατημέλη. Ήμουν πρόσφατα στην Αυστρία και συζήτησα με Αυστριακούς και μου έλεγαν όλοι αν θέλεις μεγάλης έκτασης ανακαινήσεις πρέπει να λύσεις το πρόβλημα ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις με ένα μεγάλο συγκρότημα για παράδειγμα Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, ένας αρκεί να, για να μπλοκάρει μια καλή απόφαση, επειδή περίτε ομοφωνία. Τι σημαίνει αυτό? απλούστεροι κανόνες προς όλες τις κατευθύνσεις. Το ίδιο για την ε, φορολογική, δημοσιονομική, πολιτική. Όλοι γνωρίζουμε ότι η είναι μια εθνική υπόθεση. Όμως, όταν είναι τόσο φθηνό το πετρέλαιο ή το αέριο, τότε δεν υπάρχει κίνητρο ανακαίνησης. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να καταστρώσουμε έναν οδικό χάρτη για τα κτίρια και επί της ουσίας μετά να δούμε την έκθεση, να την τροποποιήσουμε αν χρειαστεί. Και το δεύτερο θέμα, επί το οποίο είχα κάποιες απορίες, είναι το εξή. Θα συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι, οι εμπλεκόμενοι. Α πούμε, η Δανία έχει συνταξιδωτικά ταμεία, τα οποία πληρώνουν για τη δημιουργία σχετικών χρηματοδοτικών ταμείων για το περιβάλλον. Θα χρειαζόμαστε εδώ υπηρεσίες μιας στάσης στο οποίο μας θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή και ανακαίνιση κτηρίων. Να δω λοιπόν τι έχουμε, τι λείπει κλπ. Δεν είναι μόνο οι τεχνολογίες, είναι και ένα θέμα επιχειρηματικού μοντέλου. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Οπότε ένα ερώτημα είναι, δεν θα έπρεπε να οργανώσουμε ένα φόρουμ εμπλεκομένων σχετικά με την ανακαίνιση των εφισταμένων κτηρίων. Πλάι δηλαδή στον ε, μακροπρόθεσμο αυτό οδικό χάρτη. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος κ. Ζουμπίκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπέντσεν ε, για αυτό το σχέδιο έκθεσης ε, γιατί πρόκειται για μία από τις εκθέσεις οι οποίες αποτελούν μία από τις σημαντικές εκθέσεις οι οποίες δηλαδή μπορούν να συμβάλλουν στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Αν λάβουμε δηλαδή υπόψη ότι έχουμε 140 εκατομμύρια κτίρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, αποφασίσουμε να υπάρξει μια ανακαίνιση ενό συγκεκριμένου ποσοστού αυτών, πραγματικά μπορούμε να καταπολεμήσουμε και την ανεργία. Αλλά για κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε βέβαια και την ε, διεύρυνση των δεξιοτήτων των αρχιτεκτόνων και όλων των τεχνικών που θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Επίση, χρειαζόμαστε νέου τρόπου για το return on investment, δηλαδή τρόπου υπολογισμού για του ιδιοκτήτε αυτών των κτηρίων προκειμένου να μπορούν να υπολογίζουν δηλαδή το ποια θα είναι τελικά η ε, απόσβεση, ποια θα είναι η απόδοση της επένδυσης που θα κάνουν. Να μπορούν δηλαδή να βλέπουν απτά ότι πραγματικά αν προβούν σε μια τέτοια επένδυση μπορούν μέσα σε συγκεκριμένο αριθμό ετών να επιτύχουν πολύ σημαντική ε, απόδοση της επένδυσης αυτής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, συμβάλλουμε και σε αυτούς τους τομείς της ε, επένδυσης, δηλαδή των επενδύσεων και της χρηματοδότησης καθώς και της διεύθυνσης των δεξιοτήτων. Από εκεί και μετά φυσικά και θα πρέπει να ε, έχουμε πάντα κατά νου το να μην επιβαρύνουμε με ε, συμπληρωματικά βάρη τους ε, πολίτες μας. Άρα λοιπόν και στο εφορολογικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε τα ποσοστά απόσβεσης φορολογικά έτσι ώστε η χρηματοδότηση αυτών των μέτρων ενεργειακής απόδοση να είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτή και να δημιουργεί ταυτόχρονα και κίνητρα τα οποία θα προωθούν τέτοιου είδους ε, επενδύσεις, για παράδειγμα μέσω ακριβώς ε, των κατάλληλων φορολογικών κινήτρων ε, για υψηλότερα ποσοστά απόσβεση. Κάτι τέτοιο δηλαδή θα είχε πολύ σημαντικό όφελο και για το σύνολο των κοινωνιών αλλά και για επιμέρους πολίτες και νομίζω πως είναι σημαντικό. Τώρα σε ό,τι αφορά την σύνδεση τη συνδεσιμότητα σε επίπεδο ηλεκτρική ενέργεια, η κινητικότητα φυσικά αποτελεί σημαντικό πρόβλημα εδώ γιατί ε, δεν είναι μόνο οι πρίζες ε, σημαντικές ε, για κάθε διαμέρισμα, αλλά από εκεί και μετά το σύνολο του έξυπνου δικτύου, όπως λέγεται το Intelligent Grid. Εάν έχουμε δηλαδή ένα αυτο, ε, αυτοκίνητο με ε, μια μπαταρία που ζυγίζει 500 κιλά, βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα πόση ώρα χρειάζεται για να φορτιστεί όταν είναι για παράδειγμα μια από τι 500 κιλοβάτ. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μα. Έχετε δίκιο. Το πιο σημαντικό κίνητρο θα ήταν η εξοικονόμηση χρημάτων, χρήματα στην τσέπη μας. Τουλάχιστον στο μέλλον. Αν μπορούσαμε να πούμε κάτι σχετικό στην έκθεση, αν μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, ε, αυτό θα αποτελούσε για τους πολίτες μας ένα εξαιρετικό κίνητρο. Μήπως λοιπόν πρέπει να πούμε κάτι περισσότερο προκειμένου στην έκθεση. Κύριε Βέντερ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική από Γενική Ενέργειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Μπένσον για την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ τους Σκιώδης και την συζήτηση. Η Κομισιόν με πολύ χαρά θα σας γνωστοποιήσει λεπτομερή στοιχεία πώς ωφελείται δηλαδή ο κατανοητής από τα μέτρα αυτά ενεργειακής απόδοσης. Πώς προείπα το πακέτο ενεργειακής απόδοσης και χαίρομαι πολύ που μαζί ουσιαστικά συντάσσουμε μια καλή έκθεση. Δύο παρατηρήσεις επί των σχολείων των βουλευτών. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική για την ανακαίνιση. Είναι καλό τα κρατημέλη να ξέρουν ότι υπάρχει μια μακροπρόθεσμη προοπτική, πιο μακροπρόθεσμη σε σχέση με την σημερινή στρατηγική. Δεύτερον, ως προς την χρηματοδότηση, συμφωνώ. Χρειαζόμαστε επενδύσεις, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με μεγάλα κεφάλαια, όμως τομέας προτεραιότητας είναι τα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεργαζόμαστε εκεί με τη Γενική Διεθνή Ρέγγιο. 17 δις θα δαπανηθούν από το 2014 στο 2017 για έργα ενεργειακής απόδοσης διπλάσια από την προηγούμενη περίοδο. Όμως, η ανάλυση γίνεται κατά χώρα για να δούμε δηλαδή πόσα χρήματα προφήθηκαν, σε ποια χώρα, πόσο χρησιμοποιήθηκαν, πόσο αξιοποιήθηκαν. Ε, η DG Regio δεν έχει κάποιον περιορισμό, αλλά να δούμε τι είναι στη Ρουμανία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πάντως ε, θα κινηθούμε με γνώμονα τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ταμείο ε, Συνοχής. Έχουμε καλά παραδείγματα από διάφορες ε, χώρες, ας πούμε στην κοινωνική κατοικία, στη Γαλλία, στο Παρίσι, εμπροκειμένου, όπου πολλά κονδύλια επενδύθηκαν σε αυτούς τους μηχανισμούς που ενισχύουν την κοινωνική κατοικία. Τέταρτον, κάτι σημαντικό και προκειμένου χάρηκα που άκουσα τους βουλευτές να το σχολιάζουν είναι η σταθμή φόρτισης που προτείνουμε στη σχετική οδηγία. Ένα νέο στοιχείο προκειμένου. Η ηλεκτροκίνητη κινητικότητα είναι σίγουρα προτεραιότητα. Πρέπει να είναι προτεραιότητα για τα κρατημέλη και την Κομισιόν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το υλοποιήσουμε, αλλά δεν θέλω να καταλήξουμε σε ένα πρόβλημα κότα και αυγού. Αν δεν έχετε αυτοκίνητα δεν χρειάζεται το σταθμό φόρτισης ε, και αντιστρόφως όμως εμείς θέλουμε να προαγάγουμε την ηλεκτροκινητική κινητικότητα μέσω ακριβώς σταθμών φόρτισης σε κατοικίες και γραφεία σε επαγγελματικούς χώρους. Υπάρχει ένα κόστος φυσικά. Αν όμως δείτε το κόστος ενός σταθμού φόρτισης, μιλάμε για περίπου 2.500 ευρώ σε κτίρια εκτός κατοικιών. Ας πούμε ένας χώρος γραφείων με 10 θέσεις στάθμευσης, εκεί το κόστος της ανακαίνησης είναι πολύ υψηλότερο και το κόστος το κόστος της εγκατάστασης θερμοφόρτησης είναι 1,5% του συνολικού κόστους ανακαίνησης του συνολικού κτηρίου. Δεν μιλάμε για πολλά λεφτά λοιπόν. Αλλά πρέπει να στείλουμε το σωστό μήνυμα, πρέπει να δώσουμε τα σωστά κίνητρα. Σύμφωνα με τα σενάρια που προωθούμε, πρέπει οι σταθμοί φόρτισης να, όλο, να συμπληρώσουν τις φυσταμένες υποδομές, γενικότερα τις ενεργειακές υποδομές. Φυσικά οι 10 θέσεις που έλεγα σε γραφείων 10 θέσει φόρτιση είναι μόνο το 10% των πραγματικών αναγκών. Αλλά είναι καλό ξεκίνημα. Η οδηγία λοιπόν δίνει το σωστό σύνθημα, το σωστό μήνυμα τόσο για κατοικίε όσο και γραφεία και άλλου χώρου. Για την ενεργειακή ένδυα. Και εδώ η ενεργειακή απόδοση μπορεί να κάνει πολλά. Τα μέτρα βελτίωση λοιπόν τη ενεργειακή απόδοση μαζί με τα κοινωνικά μέτρα. Και τα δύο χρειάζονται. Και τα δύο θα κάνουν κάτι για την κοινωνία μας. Η οδηγία λοιπόν διαπιστώνει ότι μπορούμε να βγάλουμε από την οικονομική ένδια 1,5 με 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Eurostat, 23 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη ζουν σε συνθήκε ενεργειακής ένδυας σήμερα. Πιστεύω λοιπόν ότι μαζί με το Κοινοβούλιο και κάποια άλλα μέτρα και σε συνάρτηση με την οδηγία, έχουμε και άλλα μέτρα φυσικά εδώ, μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα νοικοκυριά, που είναι φτωχά νοικοκυριά. Μπορούμε να λάβουμε λοιπόν μέτρα, μεταξύ άλλων, για την ενεργειακή απόδοση. Κάτι άλλο που άκουσα εδώ στην αίθουσα και είναι σημαντικό και αυτό, είναι τα σχετικά με την ψηφιοποίηση και τα διασυνδεδεμένα σπίτια. Είναι, αν θέλετε, ο της ευφυΐας των δικτύων μας και των υποδομών μας. Είτε αυτό επιτυγχάνεται με ευρυζωνικά δίκτυα, με οπτικές ίνες κλπ. Τι είναι αυτό που κάνει τα κτίρια μας πιο ευφυή και καλύτερα διασυνδεδεμένα. Και από αυτού λοιπόν δουλεύουμε και περιμένουμε προτάσεις σας. Κάτι άλλο εξίσου σημαντικό που συζητήθηκε εδώ αλλά και αλλού είναι το θέμα της υγείας και της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Πρέπει να συγκεραστούν αντιδιαμετρικά αντιθέμενες επιδιώξεις και πετήσει, αλλά το θέμα σε κάθε περίπτωση ο αέρας στο εσωτερικό των κτίριων είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει κάθε φορά που συζητούμε θέματα ενεργειακής απόδοσης. ένα τελευταίο Είμαι στη διάθεσή σα διακόπτη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρο. Κύριε Γιάννησεν, Πρόεδρε. Πρώτον, ευχαριστώ του συναδέλφου για τα σχολεία τους. Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με του κοιόδη και με όποιον άλλον βουλευτή θέλει να κουβεντιάσουμε κάποια τροπολογία. Ε, η προθεσμία καταβολής, υποβολή με τροπολογιών είναι 8 Ιουνίου. Συζήτησαμε διάφορα άρθρα σήμερα, όμως εγώ θέλω να υπογραμμίσω την πρώτη μας ανάγκη. Αποδορικά κτίρια. Αυτό είναι το διακύβευμα. Αυτό πρέπει να το δούμε μαζί με τις ανανεώσιμες, με τα θέματα διακυβέρνησης και ούτω καθεξής. Στα 27 μέλη υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές και γι' αυτό η οδηγία είναι ουδέτερη ως προς την ε, ενεργειακή ασφάλεια κλπ. Αλλά τα κρατημέλη σίγουρα πρέπει να ανασκουμποθούν. Τώρα, τα ταμεία συνοχή, τα διαρθρωτικά κλπ. έχουν πολλή δουλειά να κάνουν εδώ. Ο ρόλο του είναι σημαντικό, όμω χρειάζονται και ιδιωτικά κονδύλια. Το κάναμε όμω και αυτό. Σήμερα υπογραμμίζω για μια φορά ότι μπροστά μα έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να υποβάλουμε μια πρόταση που θα έχει αμέριστη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι. Αυτό αποτελεί ευθύνη μας. Όμως το Συμβούλιο ακούω ότι θέλουν να αποδυναμώσουν την πρόταση. ενώ εμείς βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε σε λίγα χρόνια καλύτερα κτίρια, υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, λιγότερη ανεργία, γιατί ο τομέας αυτός μπορεί να δώσει δουλειά σε πολλούς ανθρώπους. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Αν έχετε κάποια ερώτηση ή σχόλιο, η υποβολή τροπολογία ως την προθεσμία. Ευχαριστώ πολύ προθεσμία υποβολή τροπολογιών 8 Ιουνίου 2017. Έχετε δύο εβδομάδες μπροστά σα, οπότε ευχαριστώ όλου τους σκιώδε, αλλά πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα τον εισηγητή μα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημείο 5. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Πατρικάη από, την, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της αεροπορίας. Σημαντικός τομέας, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο τομέας ε, συμβάλλει τα μάλα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Περίπου 5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι απασχολούνται στον κλάδο. Αμέσως και εμέσως. Η αξία του τομέα είναι περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κομισιόν τέλη του 2015 ενέκρινε μια στρατηγική για την αεροπορία στην Ευρώπη. Εκεί είχαμε εγκρίνει και ψήφισμα το οποίο ε, ενεκρίθη πριν από μερικούς μήνες και όπου καταδεικνύουμε τη σύνδεση μεταξύ αεροπορίας και διαστήματος. Μας φαίνεται τώρα βεβαίως ε, προφανές, αλλά έτσι είναι. Γιατί αξιοποιούμε και δίκτυα όπως ο έγνος, δίκτυα δορυφόρων, έγνος και τον Γκαλιλαίο. Πολύ ωραία. Ξεκινούμε. Κύριε Πατρικ Κάιλ, κύριε Διευθυντά, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ξεκινούμε με τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Αποτελεί τιμή μου το να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω τις απόψεις μας σχετικά με τη συμμετοχή μας ή τη συμβολή μας στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Θα ξεκινήσω ε, κάνοντας σας μια πολύ γενική περιγραφή της αποστολής του ΕΑΣΑ. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να επιτύχουμε το υψηλότερο δυνατό κοινό επίπεδο ε, προστασίας της ασφάλειας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ γενικόλογη λοιπόν ε, πρόταση αυτή, αλλά ε, καλύπτει και τους πολίτες, όσους μάλλον μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι μετακινούνται σε άλλες χώρες, στην Κίνα και αλλού, όχι μόνο σε Boeing, αλλά και σε Airbus και σε άλλα αεροσκάφη, σε άλλους τύπους αεροσκαφών. Κάτι που θα ήθελα να αναφέρω ε, είναι ότι στην εντολή μας ε, περιλαμβάνεται και το ε, υψηλότερο κοινό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Δηλαδή όταν εξετάζουμε για παράδειγμα κινητήρες αεροσκαφών πάντοτε εξετάζουμε ακριβώς και περιβαλλοντικά, περιβαλλοντικές πτυχές ώστε να διασφαλίζουμε ότι συμμορφώνονται με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Πιστοποιούμε ταυτόχρονα όλα τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί δηλαδή να υπάρχουν 28 διαφορετικές πιστοποιήσεις σε 28 διαφορετικά κράτη-μέλη, έτσι όπως δηλαδή γινόταν στο παρελθόν, εμείς άπαξ δίνουμε μια πιστοποίηση ασφαλεία σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που κυκλοφορούν εδώ της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Πράγμα το οποίο βέβαια συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ακριβώ τη ε, ε, της κοινή αυτής αγοράς ε, αεροπορίας και την υποστήριξη της ε, βιομηχανίας μας. Επίσης αναφέρω εδώ εντός αγγυλών τον στόχο του να ε, διασφαλίσουμε την ανάπτυξη αν θέλετε σύνταξη ευρωπαϊκών προτύπων Ασφαλείας για τα σχετικά προϊόντα. Και έχω βάλει αυτή την αναφορά εδώ σε αγγελές γιατί δεν αναφέρεται ρητά με αυτόν τον τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά ε, για παράδειγμα, ο αντίστοιχο οργανισμό ε, αναφέρει ότι θα ε, πρέπει να ο αντίστοιχο οργανισμό των ΗΠΑ θα πρέπει να προωθήσει την ηγετική θέση τη αεροπορία των ΗΠΑ στον κόσμο και ε, κατά αυτόν τον τρόπο και εμεί αντιλαμβανόμαστε ε, αντίστοιχα τη δική μα αποστολή και θα σα πω πώ ακριβώ προωθούμε τα προϊόντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα, δημιουργηθήκαμε πριν από 15 χρόνια, είμαστε 800 άτομα προσωπικό, έχουμε την έδρα μα στην Κολονία και έχουμε 32 κράτη-μέλη, δηλαδή 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 4 κράτη-μέλη ε, που έχουν υπογράψει μια συμφωνία σύνδεσης, δηλαδή η Ελβετία, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το ε, Λίχτενσταρ είναι τέσσερις αυτές τις χώρες. Τώρα, κάτι που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι το 70% ε, των δικών μας δαπανών του προβλογισμό μας καλύπτεται από τη βιομηχανία. Δηλαδή 96 εκατομμύρια ευρώ το 2016, 39 εκατομμύρια ευρώ από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 7 εκατομμύρια ευρώ από τις ε, τρίτες αυτές χώρες που σας ανέφερα, αλλά και κάποια ε, συγγραμματοδοτούμετα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, το 70% της χρηματοδότησης μας προέρχεται από τον κλάδο, από τη βιομηχανία. Και εμείς ε, ε επιλαμβανόμαστε μόνο ε, ε, ρυθμιστικού χαρακτήρα ζητημάτων, ε, δηλαδή ε, καονιστική εποπτεία και ούτω καθεξής. Ε, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο σε ΑΖ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει ε, ε, έλλειψη των απαραίτητων πόρων και βέβαια περικοπές των σχετικών προϋπολογισμών. Πράγμα το οποίο μερικές φορές είναι απογοητευτικό, γιατί παρότι η βιομηχανία χρηματοδοτεί το 70% των πόρων μας, και παρότι η βιομηχανία αξιώνει περισσότερα κονδύλια που θα πρέπει να επενδύονται στα προγράμματα του, ε, παρόλα αυτά ε, μας επηρεάζουν βέβαια οι περικοπές ε, του προεπλογισμού αλλά και του προσωπικού από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τώρα ε, προσπαθούμε να κατευθυνθούμε προ τα ε, νέα πρότυπα, επιχειρηματικά πρότυπα, δηλαδή ε, επιχειρήσεις οι οποίε έχουν την έδρα εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επιχειρήσει που είναι και ευρωπαϊκέ και αμερικανικέ ή από την άλλη πλευρά και ένα μοντέλο ε, επιχειρήσεων ε, οι οποίε, για παράδειγμα έχουν την έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, κατασκευάζουν τμήμα των προϊόντων του, για παράδειγμα των αεροσκαφών του στην Κίνα ή αλλού. τώρα, προσπαθούμε να, να, να εξετάσουμε τους κίνδυνους ε, που περιέχει η, σύγχρονη εξέλιξη της, του κλάδου μας, για παράδειγμα η κυβερνοασφάλεια. Και εδώ θέλω να σας τονίσω ακριβώς τη σχέση μεταξύ ε, των κινδύνων ε, της εσωτερικής ασφάλειας ε, και της εξωτερικής ασφάλειας, του safety και του security. Και εδώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα του τι προτίθεται να κάνει, τι προτίθεται να κάνουν οι ΗΠΑ ό,τι αφορά την απαγόρευση των λάπτοπ από τους επιβάτες δηλαδή στις ε, εκεί. Και από την άλλη πλευρά να σα πω ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με έναν κλάδο ο οποίο εξελίσσεται ταχύτητα. Έχουμε για παράδειγμα τα μη επανδρομένα αυτά αεροσκάφη, τα drones ε, δηλαδή, που έχουν αρχίσει πλέον να εξαπλώνονται στην αγορά και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις νέες τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε ε, την βιομηχανία μα. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν θα επικεντρωθώ σε δύο ζητήματα στο πλαίσιο τη παρουσίασή μου. Το πρώτο από αυτά είναι πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία μα ειδικότερα στο πλαίσιο της διεθνούς αγοράς και δεύτερο ζήτημα πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε έτσι ώστε να υποστηρίζουμε την ε, εισαγωγή ε, νέων τεχνολογιών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρώτο ζήτημα, ε, διεθνή παρουσία δηλαδή, το 80% των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί, όταν κανείς καταχωρεί ένα, καταχωρεί ένα αεροσκάφο σε ένα κράτο θα πρέπει το λόγο κράτο, όχι κράτος μέλο, συγγνώμη, ένα θα πρέπει να πιστοποιήσει τον λόγο αεροσκάφο. Δηλαδή αν η Airbus πωλήσει ένα αεροσκάφο στο Βιετνάμ, τότε το Βιετνάμ είναι υποχρεωμένο να πιστοποιήσει τον λόγο αεροσκάφο. Και αυτό σημαίνει φυσικά ότι για μία σειρά από αυτές τις χώρες πρόκειται για μία διοικητικού ε, ε, χαρακτήρα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως ε, έχει γίνει μια σειρα απο αυτέ τι χώρε προκειται για μια διοικητικου χαρακτηρα δηλαδη ουτω η αλλως εχει γινει μια σχετικη αξιολογηση εμεί δεν έχουμε την τεχνική δυνατότητα, την ευρυγνωμοσύνη για να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτή η πιστοποίηση που έχει ήδη δοθεί είναι η σωστή ή όχι. Αλλά σε κάποιες χώρες ουσιαστικά τώρα ε, γίνονται όλο ένα και περισσότεροι έλεγχοι και αφισβήτηση δηλαδή των πιστοποιητικών, ε, τη πιστοποίηση από την πλευρά της ΕΑΣΑ. Άρα λοιπόν θα πρέπει εδώ να υπάρξει υποστήριξη ούτως ώστε να μπορούν οι εθνικές, μας αρχές, οι εθνικές αρχές να πιστοποιούν τα προϊόντα μας. Ε, τι προσπαθούμε να κάνουμε με αυτό έχουμε δημιουργήσει 120 συνεργασίε εδώ, συμφωνίε συνεργασία, οι οποίε προβλέπουν το πώ θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με αυτέ τι τρίτε χώρε και επίση υποστηρίζουμε ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τριών ε, διμερών ε, συμφωνιών, δηλαδή αμοιβαία αναγνώριση, συγκεκριμένα με τι Ηνωμένε Πολιτείε, τον Καναδά και την Βραζιλία. Από εκεί και μετά έχουμε τέσσερι διεθνεί μόνιμε αντιπροσωπείε που τι βλέπετε εδώ, στον Καναδά, ε, στο Μοντρεάλ δηλαδή, στη Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ε, Κίνα και στη Σιγκαπούρη και έχουμε πέντε υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα παγκόσμια κέντρα μας. Σε σύγκριση βέβαια με ε, τα 150 άτομα προσωπικό που έχει αντίστοιχη αρχή ε, της αεροπορίας δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, προσπαθούμε από την πλευρά μα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τι εξαγωγέ των ευρωπαϊκών προϊόντων. Τώρα, επιτρέψτε μου να περάσω στο τμήμα της έρευνας και της ανάπτυξης. Εάν συγκρίνουμε δηλαδή τα κονδύλια τα οποία δαπανούνται στις ΗΠΑ με αυτά που δαπανούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε στην αεροπορία, ε, διαπιστώνουμε ότι έχουμε περίπου τα ίδια επίπεδα. 900 ε, εκατομμύρια ευρώ ετησίω στις ΗΠΑ ε, και περίπου τα ίδια επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από εκεί και μετά βλέπουμε ότι ο τρόπος που δαπανώνται αυτά τα κονδύλια είναι πολύ διαφορετικός. Δηλαδή στις Ηνωμένε ε, Πολιτείε έχουμε από τη μία πλευρά το EFA και από την άλλη πλευρά την NASA, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 20 διαφορετικά προγράμματα, μεταξύ αυτών και εθνικά προγράμματα, τα οποία βέβαια ε, καλύπτουν πολύ παρόμοιες δράσεις. Εκτός αυτού διαπιστώνουμε, θα δείτε εδώ δηλαδή, η έρευνα η οποία εστιάζει στην ασφάλεια απορροφά 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίω στι ΗΠΑ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορροφά μόνο 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή λοιπόν η διάρθρωση των δαπανών επιτρέπει στι ΗΠΑ να μπορούν να είναι πολύ πιο ευέλικτε, να ανταποκριθούν ταχύτερα στι μεταβολέ. Έχουν δηλαδή ένα ερευνητικό κέντρο με 200 άτομα προσωπικά. Έχουν 13 κέντρα αριστείας ε, στα οποία μπορούν να θέτουν ερωτήματα τα οποία είναι επίγοντα και να λαμβάνουν και τις κατάλληλες απαντήσεις νομοσύνης. Και βέβαια δαπανούν πολλά κονδύλια στην αξιοποίηση των κοινοτομιών. Επίση, εκείνο που θα πρέπει να μα ανησυχεί είναι ότι άλλε χώρε όπω η Κίνα, αλλά και η Ιαπωνία και η Νότιο Κορέα επενδύουν όλο και περισσότερο και με όλο και πιο διαρθρωμένο τρόπο ακριβώς την έρευνα και την ανάπτυξη. Όταν συγκρίνουμε δηλαδή αυτές τις χώρες με εμάς, θα διαπιστώσουμε ότι ε, ο οργανισμός ΕΑΣΑ δεν έχει προϋπολογισμό ε, για αυτό το τομέα έρευνα και ανάπτυξη. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να αξιοποιούμε τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτούμε αυτές τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Και μάλιστα Προσπαθούμε να το κάνουμε με περιορισμένο τρόπο ε, σε ό,τι αφορά πολύ συγκεκριμένα ζητήματα ασφαλείας της αεροπορίας. Ε, εάν όμως προκύψει ένα κίνδυνο, όπω για παράδειγμα σήμερα στι ΗΠΑ σε ό,τι αφορά ε, μια πυρκαγιά που μπορεί να προκύψει από μπαταρίε λιθίου, οι οποίε βρίσκονται στο αμπάρι. η ξεκινάει ακριβώ τι αντίστοιχε έρευνε με το ε, με το ερευνητικό της, ε, με το, με το εργαστήριο που έχει, ενώ αντιθέτω ε, ο ΕΑΣΑ δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν έχει την υποδομή αλλά ούτε καν και τους κανόνες προμηθειών για να το πράξει. έχουμε ενταχθεί στο Horizon 2020 αλλά με πολύ περιορισμένο και κατακαιρματισμένο τρόπο. Δηλαδή ο ρόλος που παίζουμε στον τομέα της έρευνας στο πλαίσιο του Horizon 2020 είναι πολύ περιορισμένο σε σύγκριση με το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουμε και θα έπρεπε να ε, είναι και πιο οργανωμένος και δομημένος αυτός ο ρόλος μας. Τέλος, δεν υφίσταται κάποιος μηχανισμός για την αντιμετώπιση, όπως σας είπα, επιγόντων ε, ζητημάτων. Άρα λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Και γνωρίζω πως ε, η δική σας επιτροπή ε, θα παίξει εδώ καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά δηλαδή τη μελλοντική διαμόρφωση των ε, δαπανών για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει υψηλότερε δαπάνε δημόσιε σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, ειδικότερα δε εστίαση στι επενδύσει στον τομέα τη ασφάλεια τη αεροπορία, καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων χρηματοδότηση που έχουν δημιουργηθεί για αυτού του σκοπού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε την αξιοποίηση καινοτομιών μέσω τη τυποποίησή του, μέσω της καλύτερης αξιο, ευρύτερης αξιοποίησης ε, ε, των ε, καινοτομιών και μέσω της κατάλληλης προσαρμογής των κανόνων. Ε, τώρα βρισκόμαστε σε φάση αναθεώρησης του τρέχοντος κανονισμού του ΕΑΣΑ, όπου προβλέπεται ότι ο ΕΑΣΑ θα αναλάβει ε, μελλοντικά έναν συντονιστικό ρόλο σε ό,τι αφορά ακριβώ το κομμάτι τη έρευνα και τη ανάπτυξη. Επίση, στο πλαίσιο αυτή τη αναθεώρηση ε, προβλέπεται να έχει πιο ε, ορατή, πιο ισχυρή παρουσία σε διεθνέ επίπεδο. Ε, και βέβαια και για αυτά τα δύο ζητήματα είχε ταχθεί πολύ πέρα αυτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ. Your Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα θα περάσουμε στη συζήτηση. Ήσασταν σε αυτή τη θέση πόσα χρόνια? Τέσσερα. Ωραία. Και σπιπέρ. Πρώτος ομιλητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Κή για την συνοπτική εικόνα που μας έδωσε και τις προοπτικές που μας παρουσίασε ως προς το τι θα πρέπει να κάνει στο μέλλον η ο ΕΑΣ. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την πιστοποίηση, ε, αυτή την περίοδο στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών κάνουμε το ίδιο με την αρμόδια, δηλαδή Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων. Οπότε νομίζουμε πω οι προσπάθειέ σα ε, σίγουρα είναι εντυπωσιακέ, ειδικότερα δε και στον τομέα τη έρευνα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να θέσω ένα πιο κριτικού χαρακτήρα ερώτημα. Εσεί ονομάζεστε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια τη Αεροπορία. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας οργανισμός ή οργάνωση αν θέλετε η οποία ονομάζεται Eurocontrol για την ασφάλεια της αεροπορίας. Δηλαδή την ίδια ονομασία έχετε με την Eurocontrol. Η Eurocontrol έχει 41 κράτη-μέλη, εσείς, εσείς ως ΕΑΣΑ έχετε 32 κράτη-μέλη. Και ε, λέτε ότι δεν έχετε την κατάλληλη χρηματοδότηση. Δεν θα μπορούσε να είναι μια καλή ιδέα στενότερη συνεργασία μεταξύ ΕΑΣΑ και Eurocontrol και αξιοποίηση συνεργειών. Γιατί βέβαια πολλούς δεν τους ενδιαφέρει τελικά εάν κάτι λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Το ζητούμενο είναι οι εργασίες που γίνονται να είναι ρεαλιστικέ, ε, ε, να γίνονται με αποδοτικό τρόπο και χωρίς ε, επανάληψη των εργασιών. Δεύτερο ερώτημα τώρα. Είστε πολύ περήφανος για το γεγονός ότι ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξίωσε στο πλαίσιο του κανονισμού του ΕΑΣΑ να ε, προβλέπονται περισσότερα, δηλαδή να προβλέπεται ισχυρότερο ρόλο του ΕΑΣΑ. Εγώ έριξα μια ματιά σε αυτό τον αναθεωρημένο κανονισμό, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει μελλοντικά να του ανατεθεί να πιστοποιεί ε, τον εσωτερικό εξοπλισμό των αερολιμένων και μάλιστα σε όλο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού υπάρχουν ήδη πρότυπα τα οποία είναι αναγνωρισμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οποία δηλαδή εφαρμόζουν όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί χρειαζόμαστε και πάλι εδώ νέα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν είναι μια ε, περιττή γραφειοκρατία, μια τέτοια διαδικασία, η οποία ε, θα απορροφήσει κονδύλια τα οποία ακριβώ λέτε ότι δεν έχετε στη διάθεσή σα και ότι τα χρειάζεστε. Τρίτο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τα σχέδια έκτακτη ανάγκη. Δηλαδή, αν κάτι πάει στραβά εντό εισαγωγικών σε έναν ευρωπαϊκού αερολιμένα, ο ΕΑΣΑ θέλει στο μέλλον να έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει εκεί πιο άμεσα, δηλαδή δικαίωμα εποπτείας αν θέλετε των ε, αερολιμένων των κρατών μελών. Ε, μπορείτε να μου διευκρινίσετε τι ακριβώς ε, προβλέπετε εδώ, δηλαδή πόσο ε, μεγάλο θα είναι αυτό το δικαίωμα που θα λάβει ο ΕΑΣΑ, ακριβώς σε περίπτωση όπου εντοπίζει ένα πρόβλημα σε έναν αερολιμένα ενός κράτους μέλους. Ποια θα είναι τα δικαιώματα που θα έχει και πόσο θα θέλει ο ίδιος ο ΕΑΣΑ να παρεμβαίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφος Κόκλιτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ακούσαμε προηγουμένως και θα ήθελα να σας πω και εγώ δύο λόγια στα γαλλικά ενδεχομένως μια και είναι η μητρική σας γλώσσα. Γιατί θέλετε ως ΕΑΣΑ να εφαρμόσετε τα δύο τελευταία χρόνια τους ίδιους κανόνες που αφορούν τα μεγάλα αεροπλάνα, τους ίδιους κανόνες που αφορούν τα μεγάλα αεροπλάνα να εφαρμοστούν και για τα πιο μικρά αεροπλάνα. Αυτό είναι σαν να εφαρμόζαμε τους ίδιους κανόνες, ε, τους κανόνες που για τα αυτοκίνητα, να σε εφαρμόζαμε για τα ποδήλατα. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια καταστροφή αυτού του κλάδου της ευρωπαϊκής αγοράς. Και βεβαίως θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αντιδράσεις των παραγωγών γιατί έχουμε τα ελαφριά, LSA, υπερελαφριά κτλ. Ε, έχουμε αλλαγέ σε αυτέ τι κατηγορίε. Ε, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Γιατί θέλετε να κάνετε αυτέ τι αλλαγέ, Γιατί νομίζω ότι είναι κατά στην ουσία της ευρωπαϊκής παραγωγής που είναι πολύ προχωρημένη σε επίπεδο παραγωγής. Οπότε εδώ έχουμε κάποιες απορίες. Θα Θέλω λοιπόν κάποιος ευκρινίζει αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας. Δεύτερη ερώτηση. Αν εγκρίνεται, ας πούμε, για τα μικρά αεροσκάφη μέχρι 19 επιβάτες, είναι απαραίτητο οι δοκιμές να είναι τόσο ακριβές. Γιατί για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου, όχι των μεγάλων αεροσκαφών, έτσι, αλλά των μεσαίων να τα πω έτσι, νομίζω ότι κοστίζουν πάρα πολύ οι δοκιμές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Κύριε Κουέκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Πάτρικ για την παρουσία του και για την παρουσίαση. Το θέμα παραμένει ότι ο ρόλος αυτής της υπηρεσία είναι για την ασφάλεια. Και εδώ με ασφάλεια εννοούμε ότι καλύπτουμε κάποια θέματα τεχνικής φύσης που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με την ασφάλεια σε διάφορες φάσεις της πτήσης. Έχουμε επίσης και διαφορά βεβαίως μεταξύ safety και security. θέματα που δεν είναι μόνο τεχνικά βέβαια, αλλά έχουν να κάνουν και με την αστυνόμευση, αλλά το πραγματικό ερώτημα εδώ είναι το εξής. Και αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα που θέτω στο Πατρίκ. Πού αρχίζει και πού σταματάει η ασφάλεια των αερομεταφορών. Ακούσαμε, ας πούμε, για τα λάπτοπς φορητούς υπολογιστές προηγουμένως που θέλουν να απαγορεύσουν οι Αμερικανοί. Βλέπουμε τι γίνεται. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την δουλειά της υπηρεσίας με το προσωπικό και τους που έχει με την έρευνα, δηλαδή συντονισμός, δυνατότητα παρέμβασης κλπ. Γιατί η υπηρεσία ασφάλειας δεν είναι μια ερευνητική υπηρεσία. Εξαλλού έχουμε και πολλά να κάνουμε σε σχέση με την πολιτική ας πούμε, των ΗΠΑ που οδηγεί μια διάχυση, μια διάσπαση. Οπότε και εδώ τίθενται κάποια ερωτήματα. Και έχω και ένα τρίτο ερώτημα. Η αποστολή και ο ίδιος ορισμός της υπηρεσίας όπως την όρισαν δηλαδή η Ένωση και οι συνθήκες της. Είναι συμβατή και με την έρευνα και την εμπορική της αποστολή ή αυτή η εμπορική αποστολή τέλο πάντων αποζημιώνει ότι επιτρέπει τη δημιουργία συμπληρωματικών πόρων μιας να κάνουμε τον προπολογισμό της ε, Ένωσης, ο οποίος όμως επιφέρει κάποιους περισμούς όσον αφορά το προσωπικό. Υπάρχει μια απόκληση σε σχέση με τον κανονισμό του δημοσιονομικού και του καλού που αφορούν Δεν ξέρω αν τα λέω καλά, λέει ο μιλητή. Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέλω να θέσω στα τρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρο. Να προσθέσω και εγώ κάνα δύο ερωτήματα δικά μου για την ε, ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Έχετε συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί. Μία από τις πιθανές λύσεις είναι το να βελτιώσουμε το FP9, το επόμενο δηλαδή πρόγραμμα πλαίσιο. Αλλά δεν ξέρω, ίσως εδώ έχετε κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις ή συμβουλές για το τι θα πρέπει να αλλάξει, τι θα πρέπει ας πούμε να βελτιωθεί ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας. Μετά η κίνδυνη της η ψηφιακή από τον κυβερνοχώρο. Πώς θα μπορούσαμε να σας αντιμετωπίσουμε εδώ σε σχέση με το θέμα που συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Επιτρέψτε μου να τις απαντήσω χωριστά. Ο κύριο Πίπερ καταρχάς για τη σχέση μας με το Eurocontrol. Το Eurocontrol είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία για την εναρία κυκλοφορία. Εξειδικεύεται λοιπόν στην εναρία κυκλοφορία στα πλαίσια της αεροπλοείας. Και πράγματι συζητάμε τα τελευταία τέσσερα χρόνια με την Eurocontrol για το πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και να αξιοποιήσουμε τέλος πάντων αυτό το, τον όγκο και τεχνογνωσία που έχει η Eurocontrol. Έχουμε υπογράψει και πριν δύο μήνε και μια συμφωνία για το πώ θα συνεργαστούμε για να αποφύγουμε δηλαδή επικαλύψει μεταξύ ΕΑΣΑ και Eurocontrol και αυτή τη στιγμή να αναπτύσσουμε αυτό τον τεχνικό δικό χάρτη όπως τον λέμε ακριβώς για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία και να δούμε σημείο πώς θα συνεργαστούμε. Υπάρχει λοιπόν φως εδώ στο τούνελ για τη σχέση μεταξύ Eurocontrol και EASA. Τώρα για την υποδομή των αερολιμένων. Νομίζω ότι η εντολή αυτή δόθηκε το 2009 στην ΕΑΖΑ με τους αερολιμένες. Αναπτύξαμε κάποιους κανονισμούς για τους αερολιμένες μέσα σε 3-4 χρόνια και ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται παντού στην Ευρώπη. Με στόχο να ολοκληρώσουμε φέτος, στο τέλος του έτους. Βέβαια υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, άλλες όπως η Γερμανία αντιμετωπίζουν. Τώρα δεν θέλω βέβαια να επισταθώ σε λεπτομέρειες αυτού του θέματος, αλλά τώρα κατά πόσο εμείς προσθέσαμε νέες προϋποθέσεις νέα προαπαιτούμενα σε σχέση με αυτά που ήδη υπάρχουν εθνική βάση. Αυτό ισχύει, αλλά προσθέσαμε μόνο προαπαιτούμενα τα οποία αφορούσαν χώρες οι οποίες δεν είχαν δηλαδή προδιαγραφές προϋπάρχουσες για τις υποδομές των αερολιμένων. Σε κάποιες χώρες η κατάσταση πιο δύσκολη σε σχέση με κάποιες άλλες. Δηλαδή, Πρέπει να δούμε συνολικά τι γίνεται παγκοσμίω όσον αφορά την υποδομή των αερολιμένων. Τώρα για την εποπτεία και την παρέμβαση εμείς ε, δεν θα αναλάβουμε καθήκοντα εκτάκτης, εκτάκτης ανάγκης. Λέω ο κανονισμός θα πρέπει να το διασφαλίσουμε ώστε σε κάθε αερολιμένο να υπάρχει απαραίτητη οργανωτική δομή η οποία τέλο πάντων θα αναλάβει τις ε, απαραίτητες δράσεις σε περίπτωση εκτάκτης ανάγκης. Αυτό λέει ο κανονισμός και αυτό εμείς ελέγχουμε. Δηλαδή δεν παρεμβαίνουμε οι ίδιοι με εποπτεία οι παρεμβάσεις, απλά και μόνο ζητάμε ο κάθε μένας να έχει ένα δικό του σχέδιο έκτακτης ε, ανάγκης, το οποίο ισχύει για όλα βέβαια τα αεροδρόμια αυτή τη στιγμή, ώστε τα αεροδρόμια ακριβώ να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν. Ελπίζω εδώ να απάντησα στο ερώτημα σας. Τώρα στα γαλλικά θα περάσω αν σας πειράζει για την δεύτερη ερώτηση. Από τότε που ανέλαβα, δαπάνησα πολύ χρόνο στην, ε, για την μεταρρύθμιση της πιστοποίησης των μικρών αεροσκαφών. Γιατί είπατε, δαπανήσαμε υπερβολικά πολύ χρόνο και ενέργεια για την πιστοποίηση των μικρών αεροσκαφών σαν να ήταν μεγάλα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς ε, εκδώσαμε ένα φιλοπορία γενικής αεροπλοίας το οποίο έγινε δεκτό θετικά από το σύνολο του κλάδου ως ένα μείζον σημαντικό γεγονός στα πλαίσια της αεροπλοείας. Και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια πιστοποίηση για τα μικρά αεροσκάφη, η οποία είναι πολύ πιο ταχεία και λιγότερο ακριβή από ό,τι πριν πέντε χρόνια. Τώρα, για τα ultralight αεροσκάφη και τα LSA, δηλαδή τα πολύ ελαφριά τμήματα της αεροπλογίας, τα οποία πιστοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, εμείς οι ίδιοι δεν θελήσαμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτή την νομοθεσία. Δηλαδή, οι χώρες μέλη ή κάποιες χώρες μέλη προσπάθησαν να μετακινήσουν το όριο πέραν του οποίου πιστοποιούσε η ΆΣΑ. Και έγιναν συζητήσεις μεταξύ χωρομελών, κοινοβουλίου, κομισιών για αυτά τα θέματα. Πάντως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι έχουμε όλο και περισσότερες Επιχειρήσει μικρομεσαίε που προέρχονται από τον κλάδο αυτό των light αεροσκαφών, που μα ζητούν εφ' εξής, να πιστοποιούμε τα αεροσκάφη τους. Για ποιο λόγο. Επειδή κυρίως για την αμερικανική αγορά που είναι πιο μεγάλη για αυτά τα αεροσκάφη, οι Αμερικάνοι δεν έχουν αυτή την ε, ε, έννοια, τέλο αυτή την, αυτό τον όρο ultralight. Οπότε αν εξαχθούν στη ΣΥΠΑ θα πρέπει να πιστοποιούνται από την ΕΑΣΑ να σα δώσω κάποια παραδείγματα αεροσκαφών που πιστοποιήσαμε εμεί με τη νέα προσέγγιση, τη δικιά μα, έτσι πολύ πιο ευέλικτη, λιγότερο ακριβή για τη βιομηχανία κτλ. Και η οποία είχε τεράστια επιτυχία στη ΣΥΠΑ, αλλά και στι χώρε μα, επειδή ακριβώ μπορέσαμε να προσαρμοστούμε στι ανάγκε που υπάρχουν. Και επειδή ακριβώ το πιστοποιητικό ΙΑΖΑ αναγνωρίζεται στο εξωτερικό, κάτι το οποίο δεν ισχύει απαραίτητα με τα εθνικά πιστοποιητικά, με την εθνική πιστοποίηση. Ελπίζω έτσι να απάντησα στο δικό σα θέμα στο ερώτημα. Γι' αυτό που λέγεται τώρα ο κ. Πού αρχίζει και πού τελειώνει η ασφάλεια, η οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν ένα καλό ορισμό λέγοντα ότι η ασφάλεια μια πτήση είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη πτήση τη ίδια, Δηλαδή συμβάλλει η πτήση στην ίδια τη διεξαγωγή της πτήση. Θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή έναν τρομοκράτη ή ένα τρελό πάντων πάνω στο αεροπλάνο και δυστυχώ έχουμε όλο και περισσότερου. Όχι τρομοκράτε, τρελού ανισόρροπου πάνω στα αεροσκάφη, οι οποίοι αρχίζουν να να τσακώνονται με του άλλου επιβάτε ή αρχίζουν να επιτίθενται, α πούμε, στο προσωπικό. Αυτό είναι ένα θέμα ασφάλεια, επειδή έχουμε εδώ μία επίθεση με μία πρόθεση για σωματική βλάβη και το οποίο έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την ίδια ασφάλεια της πτήσης επειδή το πλήρωμα έχει άλλα καθήκοντα και όχι να αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν. Ε, εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση. Αλλά αυτό που είναι σαφές και το βλέπουμε σήμερα στην απαγόρευση των λάπτοπ στην καμπίνα να μην ένα θέμα security στην ουσία συμβάλλουμε στο, στην ασφάλεια και μάλιστα τη στιγμή που δεν έχουμε πυροσβεστήρες μέσα στα αεροσκάφη. Προσπαθούμε πάντως αυτά τα θέματα να μην είναι το ένα εις βάρος του άλλου. Γιατί βεβαίως αυτή είναι η μας άποψη, οι Αμερικανοί βεβαίως έχουν άλλη άποψη για το security ας πούμε και το safety. Οπότε εμείς προσπαθούμε έτσι να συνδυάσουμε τα δύο και να δούμε ακριβώς πού θα θέσουμε τον πύχιο στον αφορά την όλη ασφαλεία του, της πτήσης. Τώρα για την έρευνα. απαντώντας ε, στο ερώτημα του Προέδρου για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Καταρχάς χρειαζόμαστε περισσότερο συντονισμό για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πτήσεων. Δηλαδή, ε, για το οποία δεν έχουμε ένα τελικό προϊόν. Όλη η πολιτική έρευνα της Ένωσης χαράχτηκε με στόχο στη χρηματοδότηση τη βιομηχανία ακριβώ για να χρηματοδοτήσουμε νέα και κοινοτόμα ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτό είναι λογικό. Όμως αυτό γίνεται ει βάρο της έρευνα, η οποία δεν σχετίζεται με προϊόντα και την οποία θα πρέπει να κάνουμε ανεξάρτητη έρευνα. Έρευνα, ας πούμε, για το πότε αναφλέγονται οι μπαταρίες ας πούμε, των ε, φορητών υπολογιστών. Ε, δεν πρέπει να την κάνει η σε αυτή την έρμα, πρέπει να την κάνει η Ένωση. Είχαμε ας πούμε, μελέτες ε, για το θέμα ας πούμε, των κινητών. Ξέρετε ότι σας ζητάμε να σβήσετε το κινητό σας. Επειδή είχαμε μελέτες σε σχέση με τις παρεμβολές και άλλα στοιχεία τα οποία έγιναν αποκλειστικά στη ΣΥΠΑ. Επειδή σήμερα δεν υπάρχουν βιομηχανοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να επενδύσουν επειδή ακριβώ δεν υπάρχει τελικό προϊόν. Υπάρχουν λοιπόν θέματα ή προϊόντα για τα οποία θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα χωρί να υπάρχει τελικό βιομηχανικό προϊόν. Να χρηματίσουμε λοιπόν την έρευνα με κέντρα ερευνητικά, με πανεπιστήμια κλπ. Προτείνουμε λοιπόν εμεί να καθορίσουμε τα μεγάλα θέματα ασφάλεια των αερομεταφορών, ιδιαίτερα για αυτά τα ζητήματα. Εδώ η βιομηχανία, οι κατασκευαστέ θα μα βοηθήσουν από τα πρώτα στάδια, από την έρευνα και θα φροντίσουν τα προϊόντα που αναπτύσσουν να μπορούν να πιστοποιούνται από εμά. Γιατί πιστοποίηση χρειάζεται σίγουρα. Άρα συνεργαζόμαστε με την βιομηχανία προκειμένου και τέλο. πιστεύω ότι σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε κέντρα τεχνική αριστεία στην Ευρώπη. Στι ΗΠΑ έχουν 13 τέτοια κέντρα την τύχη να εργάζομαι σε ένα από αυτά. Η αρχή είναι εξαιρετικά απλή. Έχουμε ένα κέντρο αριστείας για παράδειγμα για τα κριτικά, ένα άλλο κέντρο για την αυτοματοποίηση, για τις παρεμβολές και ούτω καθεξής. Και κάθε φορά που προκύπτει μια κατεπίγουσα ανάγκη ή πρέπει να προκύπτει ένας διαγωνισμός ο οποίος θα μπορούσε να κρατήσει δύο χρόνια, τότε δίνεται η σύμβαση απευθεία, να ανατίθεται απευθεία σε αυτό το κέντρο ή σε ένα πανεπιστήμιο. Γι' αυτό θα αξίζει και εμεί να επενδύσουμε σε κάτι παρόμοιο στην Ευρώπη. Αν κατακλείδει και πάντα σε σχέση με την ερώτηση του κ. Ρικέ, το εμπορικό κομμάτι. Πολλέ φορέ μα ρωτούν πώ θα παραμείνετε ανεξάρτητοι ενώ σα πληρώνει η βιομηχανία. Ναι, Όντω, αλλά μας πληρώνει μια βιομηχανία αλλά και ο ανταγωνισμό της. Αυτό είναι η εγγύηση της ανεξαρτησία μας. Κάθε φορά που αντιμετωπίσαμε δυσκολίες επιθεμάτων ασφαλείας σε καμία περίπτωση δεν μας επηρέασαν εμπορικά ή άλλου χαρακτήρα επιχειρήματα. Αυτό το είδαμε στην πράξη. Αυτή είναι η εγγύηση. Και αυτό έγινε σε συνεργασία με τη βιομηχανία και τον ανταγωνισμό. Μάλιστα θα λέω ότι είναι προϋπόθεση ε, για να παραμείνουμε ανεξάρτητοι. Τώρα, ο κίνδυνος ε, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, το ηλεκτρονικό έγκλημα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να γνωρίζουμε, να έχουμε επίγνωση πραγματικής κατάστασης και να είμαστε έτοιμοι. Χρειάζεται επίγνωση και ετοιμότητα επίγνωση του ότι κάποιοι είναι έτοιμοι να πλήξουν τα συστήματά μας, τα συστήματα της αεροπορίας και ετοιμότητα σημαίνει ότι κάθε εμπλεκόμενος στον τομέα της αεροπορίας, της αεροπλοείας γενικότερα, έχει ένα σύστημα διαχείρισης της δικής του ασφάλειας κατά επιθέσεων. Αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Όλοι πρέπει να συμμετάσχουν. Αυτό είναι ο πρώτο πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, ανταλλαγή στοιχείων. Ο κόσμος μας αλλάζει ταχύτατα και ο κίνδυνος επιθέσεων, ηλεκτρονικών επιθέσεων είναι υψηλός. Πρέπει λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους, τις επιθέσεις, τις λύσεις που προτείνουμε για την αντιμετώπιση τέτοιων επιθέσεων. Εργαζόμεθα και στους δύο πυλώνες, έτσι ώστε όλοι λοιπόν, όπως προείπα, να έχουν ένα σύστημα σε εγρήγορση, αλλά και κυρίω κυρίως να έχουν επίγνωση των κινδύνων. Και σε κάθε διάσκεψη, συνέδριο, εξηγούμε τους κινδύνους, τους λέμε αυτή παιδιά είναι κίνδυνοι και ως προς το δεύτερο, επαναλαμβάνω, δημιουργούμε ένα δίκτυο εμπλεκομένων που αντελάσσουν στοιχεία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τους κινδύνους των κυβερνοχωρών. Οπότε παιδί με και στα δύο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσει σα. Ίσως το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ. Είναι πολύ σημαντικό κέντρο. Δεξάγει έρευνα προσανατολισμένη, εστιασμένη σε συγκεκριμένα έργα. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν εδώ να βοηθήσει. Πολύ ωραία, ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Πατρίκ Κάι. Με συγχωρείτε που δεν προέφερα σωστά το όνομά σα, Αλλά σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την εισήγηση και τι απαντήσει και τα σχόλιά σα. Και τώρα, σημείο υπαρθμόν 6. Ανταλλαγή απόψεων Αυτά για το 6 λοιπόν, αντιλέγει απόψε με τον κύριο Πατρική, διευθυντή του ΕΑΖΑ. Έχουμε να συζητήσουμε και τα θέματα των εκπομπών αεροσκαφών τρίτων χωρών στο πλαίσιο του ETS. Η συζήτηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του έτους. Υπάρχει προθεσμία λοιπόν και εδώ διότι η τρέχουσα εφισταμένη νομοθεσία παρέχει εξαιρέσεις απαλλαγές μόνο μέχρι τα τέλη του 2017. Ο σητής, ο κ. Λάγκεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επειδή έχουμε τόσους πολλού παρεμπισκόμενου, ε, θα είμαι σύντομος. Ε, όλοι θα έχετε ούτως ή άλλω ε, διαβάσει το κείμενο και τη μεταφρασή του. Όπως είπε ο Πρόεδρος, εδώ πρόκειται για έναν κανονισμό για την τροποποίηση της οδηγίας σε ό,τι αφορά το σύστημα τη εμπορία εκπομπών στον τομέα της αεροπορίας. Η Γιούλη Γκέλεγκ από την Επιτροπή ΕΜΒ είναι η κυρία εισηγήτρια και μετά ε, η Επιτροπή Μεταφορών και η δική μας η ίτρε καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί αυτής της έκθεσης. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ε, μία πρόταση η οποία, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, ε, γενικά ε, βρίσκει τη συμφωνία όλων, ε, δηλαδή και των σχεδόν εισηγητών σε εκείνη την Επιτροπή αλλά και τη άλλη Επιτροπή. Και εμεί εδώ είμαστε σύμφωνοι. Δηλαδή, το σύστημα εμπορίου εκπομπών το οποίο άρχισε να ισχύει από το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τροποποιήθηκε το 2014 λόγω ακριβώ επιπτώσεων που είχαν ω αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, αποφασίστηκε τώρα ότι οι διεθνείς κανόνες και οι διεθνείς διαπραγματεύσεις που έγιναν προκειμένου να μην υπάρξει ένα μονομερές ε, μειονέκτημα αν μόνο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο τομέα της αεροπορίας αποφασίστηκε να ε, ε, παραταθεί το καθεστώς εξαίρεσης του, του τομέα της αεροπορίας και επίσης η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας έθεσε το στόχο Ε, να ε, σταθεροποιήσει τις ε, διεθνείς εκπομπές από την πλευρά των αεροσκαφών στα επίπεδα του 2020 και να ξεκινήσει την χρησιμοποίηση ή την εφαρμογή ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών από το 2021 και μετά. Αυτό το νέο σύστημα ε, με την ονομασία Κόρσια που αναφέρεται δηλαδή στην ε, μείωση των ε, δαπανών και την περισσότερη αποτελεσματικότητα τομέα της αεροπορίας γίνονται κάποιες προτάσεις από την πλευρά της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την παράταση του καθεστώτος εξαίρεσης για το τομέα της αεροπορίας το οποίο καθεστώς εκπνέει το 2017 και γι' αυτό είναι επίγουσα η κατάστασή μας. Ε, και εδώ λέμε συγκεκριμένα δηλαδή παράταση για τις ε, περιπτώσεις εκείνες των επιχειρήσεων που έχουν ε, εκπομπές έως χιλιών τόνων. Δηλαδή εδώ προτείνουμε η Επιτροπή να αναλάβει την υποχρέωση να ενημερώνει το Κοινοβουλίο και τον Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην αιτία αγορά και προβλέπουμε επίσης το να αναλάβει το δικαίωμα υιοθέτηση σε κατεξοδότηση πράξη η Επιτροπή, στο πλαίσιο βέβαια τη διαδικασία συνένεσή μα σε ό,τι αφορά ακριβώς την θέσπιση αυτής της ε, παράταση τη εξαίρεση. Από εκεί και μετά η, το ποσοστό της μείωσης, ε, δηλαδή γραμμικής μείωσης κατά 1,74% παραμένει ως έχει και από εκεί και μετά βέβαια η προθεσμία είναι σύντομη ούτως ώστε να προλάβουμε να κάνουμε τα πράγματα στο σωστό χρόνο. Δηλαδή το, η γραμματεία πρότεινε μετά την εξέταση σήμερα της έκθεσης 1η ε, Ιουνίου, Παρασκευή δηλαδή το μεσημέρι να έχουμε την, ε, την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και να την υιοθετήσουμε 21 έκτου. Ε, στην Επιτροπή μας για να ακολουθήσει μεταθέτηση και από την ε, ΕΝΒ. Εμείς ε, λοιπόν στην πρότασή μας υποστηρίζουμε τα όσα από την Επιτροπή, αλλά έχουμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις, κυρίως διατύπωσης με 8 συνολικά τροπολογίες. Οι δύο σημαντικότερες από αυτές τις τροπολογίες είναι ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση πρόσφατα ότι η συμπερίληψη πτήσεων σε τρίτες χώρες σε ένα χώρο, ε, σε, σε ένα αερολιμένα του ΕΟΧ δεν έρχεται σε αντίθεση με το διεθνέ δίκαιο. Παρόλα αυτά, μια τέτοια ρύθμιση θα οδηγούσε σε πολύ σημαντικέ ε, διαμάχε με τη Ρωσία και άλλου ε, διεθνεί εταίρου, οπότε θέλουμε να διαγραφεί αυτό το σημείο. Δεύτερο σημαντικό, δεύτερη σημαντική τροπολογία. Θεωρούμε ότι η σταθερότητα των διεθνών συμφωνιών και η αιμονή σε αυτή τη σταθερότητα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο περιγράφει η Επιτροπή. Άρα λοιπόν πέρα από τα υποχρεώσει υποβολή τη έκθεση προτείνουμε η Επιτροπή να έχει μια συμπληρωματική υποχρέωση να μειώσει αν θέλετε λίγο τα, τον πύχη που έχει θέσει τον εαυτό τη, να μειώσει αυτά τα πρότυπα που έχει θέσει, αλλά παρόλα αυτά να παραμείνει φιλόδοξη και κατά συνέπεια να προβαίνει σε αξιολόγηση αντικτύπου μια εκτίμηση του πώς αυτό το κόρζια, αυτό το διεθνές δηλαδή σύστημα εκπομπών, ε, το οποίο θα ισχύσει από το 2021, θα, ε, πώς ε, θα εξελίσσεται λοιπόν αυτό το κόρζια και πώς θα μπορούν να συνεπάρχουν παράλληλα το δικό μας σύστημα εμπορίας και το κόρζια από το 2021. Αυτές λοιπόν είναι οι προτάσεις που κάνουμε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε και νομίζω πως οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το ζήτημα έχουν παρακολουθήσει την όλη συζήτηση. Ευχαριστώ, λέω πρόεδρο, στη Ραντεμόντε. Από του σοσιαλιστέ. Μια γενική παρατήρηση. Γιατί είναι απαραίτητο να επανέλθουμε στο θέμα των εκπομπών. Είχαμε μια αύξηση 30% από τότε στον αφορά στο 80, το 90 συγγνώμη, είχαμε και αύξηση της κυκλοφορίας. Φέτος διψήφιος ο αριθμός της αύξησης. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή και συμφωνώ με τα μέτρα της Κομισιόν που είναι φιλόδοξα να μειώσουμε δηλαδή μέχρι το 2030 30 κατά 40% αυτό που είχαμε από το 90. Πρέπει όμως να υπάρχει σαφήνεια για τους φορείς και τους εμπλεκόμενους και πρέπει γρήγορα, γρήγορα να θεωρηθεί το κείμενο με προθεσμίες που θα μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε σε αυτά που προβλέπει το σύστημα για τις αερομεταφορές. Επίσης για την περίοδο 17-20 θα πρέπει να διατηρηθεί το τωρινό πεδίο εφαρμογής δηλαδή η πτήση στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Για την υλοποίηση τώρα του μέτρου αυτού παγκοσμίω θα πρέπει να κάνουμε μια αναβολή όσον αφορά το σύστημα ITS για την περίοδο μετά το 2020. Μέχρι δηλαδή να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με την φύση και το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας και των προθέσεων των διεθνών μας εταίρων. Πάντως είναι σημαντικό να είναι έτοιμη η Ένωση και οι χώρες για περαιτέρω αξιολόγηση του συστήματος αυτού μετά το 20. Και αυτό ακριβώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με την Κομισιόν ώστε να αντιμετωπίσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις εκπομπές από τις διεθνείς αερομεταφορές. Στηρίζω λοιπόν αυτή την γνωμοδότηση όπως έχει συνταχθεί και με τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Από πλευρά μου όμως θα κάνω κάποιες διορθώσεις ώστε να έχουμε ένα ξεκάθαρο κανονισμό και ο οποίος θα υιοθετηθεί γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου, κυρία Φύρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που είπαν ότι υπάρχουν πολύ καλά στοιχεία στην έκθεση. Εγώ είμαι ικανοποιημένη από το βάρος που δώσαμε στον τομέα της αεροπλοείας και την ανταγωνιστικότητά του. Σύμφωνα με τις προθεσμίες κλπ. Ο ΙΚΑΟ επίσης έχει κάνει πολλή δουλειά στον τομέα. Πρέπει να συγκεράσουμε την οικολογία με την οικονομία, τα κίνητρα με την ρύθμιση. Η ισορροπία είναι απολύτως απαραίτητη. Όμως υπάρχουν και πράγματα που λείπουν από την έκθεση και θα ήθελα να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Εγώ ας πούμε ταξιδεύω μέσω Ζάβεντεμ, ξέρω πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι τα αεροδρόμια για την εθνική οικονομία και την οικονομία γενικότερα. Και γι' αυτό συμφωνώ ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να συγκεράζουμε, όπως προείπα, την φροντίδα για το περιβάλλον με την ανταγωνιστικότητα της αεροπλοείας μας. Θα πρότεινα λοιπόν τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπών να επενδύονται στην έρευνα για καθαρότερο περιβάλλον. Αυτό θα ήταν μια καλή όθηση στην σχετική τεχνολογία και θα είχε ωφελήματα για ολόκληρον τον τομέα. Θα αντισταθμίζαμε έτσι και την μεταβολή του κλίματος. Εν μέρη φυσικά. Αυτό θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ γρήγορα. Μάλιστα θα δείχναμε ότι είμαστε πρωτοπόροι. Θα πιέζαμε και τον ΙΚΑΟ και άλλους ε, φορείς να κάνουν κάτι παρόμοιο. Θα περιχαίναμε λοιπόν έτσι με μία κίνηση πάρα πολλά. Πάντως πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα ανταλλαγή ε, δικαιωματών εκπομπών. Εμεί ήρθε η ώρα να πάρουμε αποφάσει. Έχει όμω μεγάλη σημασία να έχουμε και ένα εναλλακτικό σχέδιο, ένα plan B όπω λέμε φορά, στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Αυτά κατά τα άλλα θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τον εισηγητή και του ε, σκιώδε. Ευχαριστώ. Και στα Λούντα από του πράσινου Πρόεδρε. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το κλίμα απειλείται, οι εκπομπές όμως αυξάνονται. Αυτό είναι απαράδεκτο, διότι συνεχίζονται, συνεχίζονται να αυξάνονται εκπομπές παρά τη συμφωνία στο Παρίσι. Θα λέω το εξή λοιπόν, από το 2020-2021 θα πρέπει να ισχύσουν οι νέες, οι νέοι περιορισμοί Να εξαιρεθούν επίση χώρε από του περιορισμού που εφαρμόζουν την κόρσια. Πρέπει επίση να σταθμίσουμε τι επιπτώσει από το διοξείδιο του άνθρακα που είναι πολύ ψηλέ για την αεροπορία. Δεν είναι όμω μόνο το διοξείδιο του άνθρακα, είναι η αεροπλοεία γενικότερα. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν οι εκπομπέ τη αεροπλοεία με τον αντίστοιχο συντελεστή. Η αεροπλοία πρέπει να λάβει τι ευθύνε τη ε, για το πόσο επιβαρύνει τον πλανήτη, όπω όλοι οι άλλοι τομεί. Δεν πρέπει να επιτρέπει στην αεροπλοεία ούτε να παραμείνει σε ίδια επίπεδα, ούτε πολύ μάλλον βεβαίω να αυξήσει τι εκπομπέ τη. Πρέπει να προσαρμοστεί και η αεροπλοεία μετά το 2020. Τέλο. Στο πλαίσιο του ETS, του Συστήματο Συνταλλαγή Δικαιωματών Εκπομπών, συνεχίζουν να υπάρχουν κίνδυνοι που δεν αφορούν όμω την αεροπλοεία. Δηλαδή, για μια πτήση στο Χόρμπι Βρυξέλλε, το κόστο είναι περίπου 1 ευρώ. Για μια διεθνή πτήση, το κόστο είναι 5 ευρώ για κάθε επιβάτη. Το κόστος λοιπόν βλέπουμε ότι αν εισιτήριο είναι αμεληταίο. Άρα έρθει η ώρα λοιπόν, να αυξήσουμε την επιβάρυνση τη αεροπλοεία όσον αφορά τι εκπομπέ τη. Πρώτα ευχαριστώ. Ο κύριος Ηλικιώτης, από την ΚΟΑ, παρακαλώ. Πρόεδρε, ε, και για την ομάδα μας, την ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς, πρωταρχικός στόχος είναι, πρέπει να είναι η μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές δραστηριότητες για αντιμετώπιση των στόχων που θέσαμε για τις κλιματικές αλλαγές, για προστασία του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου ζητάμε λοιπόν αυστηρότερα μέτρα για τους μεγαλύτερους ρηπαντές σε όλες τις πτήσεις από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο στις πτήσεις εντός του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Δεν γίνεται να συνεχίσουν οι παρεκκλήσεις και να μην τεθούν αυστηροί κανόνες συμμόρφωσης για μία των και στις πτήσεις από και προς αεροδρόμια που βρίσκονται εντός της Ένωσης. Είναι απαράδεκτο λόγω του στόχου της αύξησης της ανταγωνιστικότητας η Ευρωπαϊκή Ένωση να θυσιάζει την προστασία της δημόσιας υγείας. Και είναι θέμα αυτό ε, ε, ε για μας να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες μας. Έπειτα, τα δωρεάν δικαιώματα πρέπει να δίνονται με αναβαθμίσεις και στοχευμένα με αυστηρά κριτήρια, ώστε να αποφορούνται μόνο όσοι έχουν πραγματική ανάγκη. Αυτό που αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να προστατήσει ώστε να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος μηχανισμός, όχι αγοροκεντρικός, ε, να στοχεύει δηλαδή στην λειτουργία της αγοράς, ε, και να εξυπηρετεί δίθεν τις ανάγκες της αγοράς, αλλά ένας μηχανισμός ο οποίος πρώτιστα και γνώμονα θα έχει τις ανάγκες της κοινωνίας, ε, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημόσια υγεία, για να μπορέσει πραγματικά να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών από τις αεροπορικές δραστηριότητες. Ε, αυτή σε γενικέ γραμμέ είναι η δική μα τοποθέτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η δεν έχει κάποια παρατήρηση, όχι. Η κυρία Λόρας Γκραφ από τη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Λάγκεν για το ότι κατέθεσε γρήγορα το σχέδιο έκθεσης και το ότι υποστήριξε εν γέννη την κατεύθυνση της Κομισιόν. Ευχαριστώ και όλους τους άλλους για τις ε, παρεμβάσεις τους. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση της Κομισιόν, ακολουθεί αυτό άλλωστε ήταν και η εντολή μας, την έγκριση στον ΙΚΑΟ προσφάτως του λεγόμενου σχήματος Κροσία, που είναι ένα παγκόσμιο σύνολο μέτρων για την αγορά με στόχο την αντιστάθμιση των εκπομπών της αεροπλογίας με ε, κάτω από τα επίπεδα του 2020. Δεν είχαμε αυτό ακριβώς στο μυαλό μας όταν ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι η εξέλιξη είναι σίγουρα καλοδεχούμενη, να μειώσουμε δηλαδή παγκοσμίω τι υπομπέ θεραπλοεία. Οπότε, είμαστε ικανοποιημένοι με το μέτρο, ιδιαίτερα μετά από το Παρίσι, γιατί όπω είπαν και πολλοί από του προλαλήσαντες αν ε, λάβουμε υπόψη μας την αύξηση της κυκλοφορίας, των πτήσεων δηλαδή, η αεροπλοεία σίγουρα πρέπει να κάνει περισσότερα για να μπορέσει να συμβάλλει στην επιτεύξη του εν στόχου, της μείωσης δηλαδή. Το πέσινο ψήφισμα ήταν φυσικά το πρώτο βήμα, όμως όπως πολλοί ήδη είπαν, έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Ωστε το COSIA να είναι επιχειρησιακά έτοιμο ήδη από το 2021 όπως είναι το σχέδιο. Δύο πτυχές θέλω να τονίσω. Πρώτον, πρέπει να συμφωνήσουμε ενό συνολού κανόνων όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή στην πράξη του μηχανισμού και ένα σύνολο κανόνων για σημαντικές πτυχές του μηχανισμού που αφορούν την διαφάνεια, του σχετικούς υπολογισμού, ε, την εσωτερική λογιστική αν θέλετε κλπ. Όλα αυτά είναι υπό διαπραγμάτευση στον ΙΚΑΟ και φυσικά είμαστε παρόντες, ε, συμμετέχω και παρακολουθώ αυτήν την διαπραγμάτευση γιατί αυτά ακριβώ τα στοιχεία είναι και τα στοιχεία κλειδιά όσον αφορά την ακαιρεότητα και την δυνατότητα εφαρμογή στην πράξη του μηχανισμού. Όταν θα φτάσουμε εκεί θα έρθει η σειρά των κρατών μελών φυσικά να τα εφαρμόσουν όλα αυτά σε εθνικό επίπεδο. Η Κομισιόν λοιπόν υπέβαλε μια πρόταση που λαμβάνει υπόψη τη όλα αυτά τα στοιχεία. Προσπαθεί επίσης να διευκολύνει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις περί το Κόρσια χάρη στο οποίο διευρύνεται και το αντικείμενο των τρέχουσων διαπραγματεύσεων. Αποφασίσαμε πάντω σε κάθε περίπτωση να υιοθετήσουμε την ίδια προσέγγιση, αυτή που είχαμε υιοθετήσει και πριν από τι περσινέ διαπραγματεύσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό, προβλέπεται αναθεώρηση της συμφωνίας από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσει κάποιο το τοπίο όσον αφορά την εφαρμογή του Κορσία από το ΙΚΑΟ και από τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάποιες άλλες σημαντικές πτυχές της πρότασής μας είναι οι εξής. Τα, τα ανέφεραν και κάποιοι από τους προλαλήσαντες. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Να εγκρίνουμε λοιπόν την πρόταση ως το τέλος του έτους σίγουρα Πρέπει συνεφώς να διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις μας, με, με με το Συμβούλιο, γιατί αλλιώς θα περιπέσουμε στην κατάσταση όπου θα αφορά ο μηχανισμός στους πάντες. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να διαχειριστεί ορθώς την κατάσταση τα επόμενα χρόνια Πρέπει να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς εξελίξεις. Πρέπει να συζητήσουμε την αναθεώρηση του ETS, ε τις ανταλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών και τι κάνουμε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Θα αρέσει να δούμε λοιπόν το μηχανισμό αναθεώρησης, να δούμε πού πηγαίνει ο ΕΚΑΟ, Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία και να παρακολουθήσουμε φυσικά και τι εξελίξει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη συμβολή στι εκπομπέ τη αεροπλοεία και πώ μπορεί η αεροπλοεία να συμμορφωθεί με του στόχου για το 2020. Χρειάζεται συνέπεια ε, συγκυρασμό, αν θέλετε, όλων αυτών των επιμέρου στόχων. Αυτά θα γίνουν, εννοείται, εν ευθέτω χρόνο, όπως προείπα, μόλις ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ΙΚΑΟ. Φυσικά δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, ούτε μπορούμε να αναφερθούμε ρητό ε, στη μία την άλλη εναλλακτική λύση. Πρέπει να διατηρήσουμε τα περιθώρια ευελιξία μα, γιατί στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ προτάσει. Αυτά προ το παρόν για του σκοπού αυτή τη πρώτη συζήτηση. Τουλάχιστον ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Τελευταίε καταληκτικέ παρατηρήσει από τον κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφους και την Επιτροπή για την υποστήριξή τους. Καλό δεύτερον, ε, ναι, από το 1990 οι εκπομπές ε, από την αεροπορία έχουν ε, προφανώς αυξηθεί, αλλά από την άλλη πλευρά έχει τριπλασιαστεί και η αεροπορία, δηλαδή ο αριθμός των πτήσεων, ειδικότερα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Ε, έχουμε λοιπόν άλλους μηχανισμούς οι οποίοι επιτυχάνουν μείωση, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά νέους κινητήρες, γιατί για παράδειγμα έχουμε μείωση των εκπομπών, άνα για παράδειγμα επιβάτη με βάση τους νέους κινητήρες, αλλά εδώ επανέρχομαι λίγο και στην ε, βασική συζήτηση που κάναμε πριν από 15 έτη, δηλαδή όταν συζητούσαμε ακριβώ την δημιουργία του συστήματο εμπειρία εκπομπών. Γιατί δεν έχει πετύχει αυτό το σύστημα, γιατί συμπληρωματικά ξανά και ξανά ε, υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία προτείνονται. Δηλαδή, αν πραγματικά είχαμε ένα αμυγέ αν θέλετε, σύστημα εμπορία εκπομπών, τα πράγματα θα ήταν πολύ εύκολα. Το 2012 συμπεριλάβαμε το τομέα τη αεροπορία εκεί ε, και ε, ήταν πραγματικά αμφιλεγόμενη αυτή η απόφαση και υπήρχε και αντίσταση από τον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα τελικά αποφασίστηκε ότι είναι αθέμητο ο ανταγωνισμό εάν δεν εφαρμοστεί ένα τέτοιο σύστημα διεθνώ και όχι μόνο για τι επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό η Επιτροπή στο πλαίσιο των φόρα των οποίων συμμετέχει να πιέσει προς την κατεύθυνση καθήτρηση ενός κοινού διεθνού συστήματος. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και βέβαια σε ό,τι αφορά το στόχο Στόχο που έχουμε θέσει σε ό,τι αφορά την κλιματική μεταβολή, διαρωτώ γιατί χρειάστηκε 1,5 χρόνο Επιτροπή μετά από τη Διεθνή Διάσκεψη στις 6 ε, Οκτωβρίου του 2016 ε, όταν δηλαδή έχουμε, έχει ήδη εκπνεύσει σχετική προθεσμία από τις 31 Δεκάτου του 2016. Με άλλα λόγια, η δική μας πρόταση είναι καθυστερημένη επειδή υπάρχει καθυστέρηση από την Επιτροπή, όχι επειδή εμείς χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για τη διαβουλεύση. Σε βάση περιπτώσει, αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα γίνει στο μέλλον και αναμένω και τις ε, τροπολογίες που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, σκιώδεις, τον ισχύτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά σας. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 1η Ιουνίου 2017. Σε τρεις μέρες δηλαδή από σήμερα. Κυρίες και κύριοι, δεν έχετε και πολύ χρόνο. Ευχαριστώ πολύ όλους. Επόμενο σημείο, αποστολή Ήτρε στο Μπερέκ, στην Ρήγα της Λετωνίας, 20-21 Απριλίου. Απολογισμός. Τρία άτομα, τρία μέλη μας πήγαν στην, στα γραφεία της Μπερέκ στη Λετωνία. Πρόκειται για τον φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Ερχών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ο Μπερέκ. Η Ήτρε επεξεργάζεται την πρόταση της Επιτροπής για τον Μπερέκ. Ο κ. Στοσινόφσκι είναι εισηγητής. Ο κ. δυστυχώς Ευτυχώς. Είναι εδώ, παρακαλώ. Σας ακούμε. Πείτε μας για την ε, επίσκεψή σας στα γραφεία του Μπερέξ στην Λετωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παρουσιάσω συντομία ε, την ε, περίληψη της επίσκεψής μας έλαβε χώρα στην κατάλληλη χρονική συγκυρία αυτή η επίσκεψη γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε μια εν μέσω μάλλον μια διαδικασία σύνταξης έκθεση ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του Μπέρεκ. Η αντιπροσωπεία μας λοιπόν αποτελούνται από τρία μέλη της Επιτροπής Ήτρε, έναν εισηγητή δηλαδή και δύο σκιώδης και Γι' αυτό πραγματικά ήρθε σε μια πολύ σωστή στιγμή. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, Γκάρδια τον ε, Μπέρεκ για, ή μάλλον το, το γραφείο του Ιτρεμ και τον Λούπε Ρίκινσον που διοργάνωσαν με τόσο αποτελεσματικό τρόπο αυτή την επίσκεψη. Είχαμε δηλαδή μια διήμερη μόνο επίσκεψη αλλά καταφέραμε στο πλαίσιο αυτής να μάθουμε όσα χρειαζόμασταν, όλα τα σημαντικά στοιχεία. και νομίζω πως θα συμφωνούσαν οι συνάδελφοι, οι άλλοι δύο συνάδελφοι που συμμετείχαν, οι οποίοι απουσιάζουν αυτή τη στιγμή, ότι δηλαδή ε, το γραφείο Μπέρεκ πραγματικά εργάζεται με υψηλότατο επαγγελματισμό. Είναι ένα μικρό γραφείο, με χαμηλό δηλαδή αριθμό προσωπικού, αλλά το έργο που επιτελεί είναι πολύ περίπλοκο και ε, θα συνεχίσει να καθίσταται όλο ένα και πιο σημαντικό και στο μέλλον. Ε, είναι πραγματικοί επαγγελματίε όσοι εργάζονται σε αυτό το γραφείο. Το σημαντικό είναι ότι ε, μάθαμε το πώ λειτουργεί σε εσωτερικό επίπεδο ο Οι παρουσιάσει που μα έκαναν ήταν πολύ ποιοτικέ Συναντηθήκαμε δηλαδή και με τον ε, πρόεδρο του Μπέρεκ, τον ε, Σεμπαστέν ε, Σεριάνο, αλλά και τον μελλοντικό πρόεδρο, τον κύριο Νούγκελ, ο οποίος μας έκανε μια παρουσίαση των, των απόψεων του Μπέρεκ. Ο κύριος Μιλάς Λοιγνάτς, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του γραφείου στη Ρήγα, ήταν σημαντικό που παρευρέθη εκεί γιατί μας έδωσε πληροφορίες άμεσες από τη δική του εμπειρία. Η συζήτηση που ακολούθησε αφορούσε την ε, νομοθεσία που συζητείται αυτή την περίοδο και η οποία θα υιοθετηθεί, αναμένεται να υιοθετηθεί τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Ε, τώρα, πώς ε, έχει η δομή του Μπέρεκ. Έχουμε τον ίδιο τον Μπέρεκ από εκεί μετά το γραφείο του. Ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα είναι το, η δημιουργία ενός συστήματος ψηφοφοριών σε ό,τι αφορά τη λήψη περίπλοκων αποφάσεων από την πλευρά του Μπέρεκ. ενώ ή ε, όλοι οι επιβεβαιωτές των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών που συμμετέχουν ε, είναι υποχρεωμένοι να ε, διατηρούν την ουδετερότητά τους. Θέσαμε κάποια ερωτήματα ως προς το προτινόμενο μοντέλο, μελλοντικό μοντέλο διάθεσης του ΜΠΕΡΕΚ, όπως δηλαδή προτείνεται από την Επιτροπή. Και αυτό που μας είπαν είναι ότι ουσιαστικά θα υπάρχει ένα διπλό σύστημα ε, διαπραγμάτευσης το οποίο ήδη λειτουργεί πολύ καλά και διασφαλίζει ένα υψηλό βαθμό απεροληψίας. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να μεταβληθεί αυτό το σύστημα διπλής διαπραγμάτευσης. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει ανετικό αντίκτυπο στις ε, ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Εγώ ως ε, εισηγητής γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με έναν ε, πολύ επαγγελματικό οργανισμό και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε κάτι το οποίο θα είχε ανετικό αντίκτυπο στη λειτουργία και στο έργο που επιτελεί. Η, η επίσκεψη, όπως σας είπα, ήρθε πραγματικά στην κατάλληλη χρονική στιγμή Ε, λάβαμε γνώση πολύ σημαντικών πληροφοριών τις οποίες ε, ε, προτιθέμεθα να συμπεριλάβουμε και στο νομοθετικό μας κείμενο. Και η Κωνσταντς Κρέλ και άλλοι είχαν συμμετέσχει Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην νομοθεσία γιατί έχουμε να κάνουμε με μια υπηρεσία η οποία είναι αρκετά ανεργή και θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Οπότε να σας ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση που μας κάνατε και ευχαριστώ για αυτή την άποψή σας ήταν δηλαδή χρήσιμο να πάμε στην ρεγιά Πρόεδρος, τώρα. Κυρία Κουντρίσκα, η κυρία Καμπεσόν η κυρία Γκέρινγκ, Ματίας και ένας άντρας συνάδελφος. Ταλούνται πέντε είχατε πάει. Στην αποστολή που θα συζητήσουμε τώρα για τη Γερμανία στο ταξίδι σα στην Πολωνία, Γερμανία. Κύριε Καπεσόν Ρουή, πείτε μα τι έγινε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. όπω ξέρετε, αύριο θα ψηφιστεί η έκθεση που αποτέλεσε το αντικείμενο της επίσκεψης που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για την προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Πήγαμε λοιπόν στο Βερολίνο, στη Γερμανία, για να δούμε το πώς λειτουργεί το ΣΔΙΔ εκεί και για να δούμε ακριβώς μια χώρα της πρόσφατης διεύρυνσης εν και του 2020. Πήγαμε στην Rolls Royce που όπως ξέρετε είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίω κινητήρων για μεγάλα αεροσκάφη και είναι μέλος και του Clean Sky που κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά ερευνητική όσον αφορά την μείωση των εκπομπών δεξιδιών άνθρακα στον τομέα αεροπλοεία. Επίση, επισκεφθήκαμε την Bombardier Transportation που είναι πρωτοπόρος στη συνδρομική τεχνολογία και είναι και ιδιωτικό μέλος του GTH και του Rail. Συζητήσαμε διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ο του ΔΙΤ για την πρόθεση της αεροπλοείας, η αξιοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων, τα ΣΔΙΤ και η συμμετοχή των πανεπιστημίων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η συμμετοχή στο Clean Sky 2 η συνεργασία με τα περιφερειακά ταμεία και τα αντίστοιχα αποτελέσματα και η υπογραφή 12 μνημονίου συνεργασίας με χώρες μέλη. Συζητήσαμε επίση θέματα έρευνας όσον αφορά προϊόντα υψηλή τεχνολογίας Μίλησαμε για τη χρηματοδότηση τη βιομηχανία και την συμβολή του ιδιωτικού τομέα στα εθνικά προγράμματα, πρόσβαση στα δεδομένα, η συμμετοχή στην έρευνα του ιδιωτικού τομέα και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπω επίση και η προετοιμασία του Κλίνσκα 3. Τη δεύτερη μέρα πήγαμε στην Πολωνία, στο Λότζ, στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο. Ένα από τα κυριότερα κέντρα, ερευνητικά κέντρα ιατρικής στη χώρα. Και εκεί συζητήσαμε για τα ζητήρια και το ρόλο τους ακριβώς στην πρόθεση της, της τεχνολογίας και της έρευνας. Είχαμε και μια παρουσίαση για θέματα υγείας από το αντίστοιχο ερευνητικό Ινστιτούτο που κάλυψε το θέμα της υγιούς ε, ζωής σε σχέση με την εξέλιξη τη δημογραφική. Μετά συζητήσαμε και την διεύρυνση της ε, συμμετοχής σε προγράμματα αέρα του ίνιν κλπ. Επίσης, συζητήσαμε τη συμμετοχή αυτών των προγραμμάτων σε σχέση με τα προγράμματα μετά το 2020. Σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση μιλήσαμε και με τους εκπροσώπους του Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου οι οποίοι μας έδωσαν μια θεσμική άποψη εικόνα και συναντήσαμε επίσης και πανεπιστημιακούς από διάφορα πανεπιστημία της ε, Πολωνίας. Συζητήσαμε και πάλι το θέμα του 2020, τι προβλήματα αντιμετωπίζει, γραφειοκρατία, καινοτομία και την έλλειψη στήριξης στην ε, στοχευμένη καινοτομία αυτή τη στιγμή. Οι συμμετέχοντες ζήσαν ακριβώς να ληφθούν ε, μέτρα ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και άλλων ερευνητικών κέντρων. Μας ζήτησαν τη συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων και μίλησαν για την διαχείριση και τη συμμετοχή ως βασικός σημείο εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων που θα εμπλέξουν και άλλους συμμετέχοντες. Αυτά ήταν κυρίως τα θέματα που συζητήσαμε, θέματα που ήταν πολύ χρήσιμα και τα οποία εντάσσονται και περιλήφθηκαν στην έκθεση που θα παρουσιάσουμε αύριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία μου, λέει ο Πρόεδρος. Είστε υπεύθυνοι για τον ορίζοντα 2020 και την αντίστοιχη έκθεση. Ελπίζω η, έκθεση, η επίσκεψη αυτή να ήταν χρήσιμη για σας και για τους σκιώδες. Και ο κύριος Τουσανόφσκι είναι υπεύθυνος για τον κανονισμό Μπέρεκ. και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η επίσκεψη στην Λετωνία. Αύριο θα τα ξαναπούμε λοιπόν συνάδελφοι, αύριο 9 η ώρα του πρωί έχουμε τους και μετά στις 10 έχουμε τις ψηφοφορίες. Οπότε θα τα ξαναπούμε στις 10. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.